Good morning to everybody. We are just waiting for the president of the court. This is all. He's appearing in one. Σε ένα-δύο λεπτά θα έρθει ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου. So, ich wünsche allen einen guten Morgen und begrüße den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes, Klaus-Heiner Lehne. Καλωσορίζω τον κύριο Λένε και επίσης και τον κύριο Λαζάρου, ο οποίος σήμερα θα μας ε, παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018. Και θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά και τον κύριο Ότιγκερ και όλους τους ε, συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά τις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου, δεν ξέρω αν έχετε κάποια παρατήρηση για την ημερήσια διάταξη ή για τα έγγραφα τα οποία σας έχουν αποσταλεί. Καμία παρατήρηση. Σήμερα η μετάφραση ε, είναι στις ε, περισσότερες γλώσσες, όχι σε όλες, στις περισσότερες και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και μετάδοση μέσω διαδικτύου, αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει μέσω διαδικτύου. Όσον αφορά τις συστάσεις των συντονιστών, τους συνεδρίασης της 26 Σεπτεμβρίου. Οι συστάσεις αυτές σας διανεμήθηκαν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις πριν από το τέλος της συνεδρίασης, οι συστάσεις αυτές εγκρίνονται, γίνονται δεκτές. Περνάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 3 της ημερήσιας διάταξης στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρο, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμη κύριε Επίτροπε Ότιγκερ, αξιότιμη εκπρόσωπο του ε, Συμβουλίου, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα βρήκατε χρόνο για το ε, ελεγκτικό συνέδριο παρότι η ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι απαιτεί τον περισσότερο από το χρόνο σας. Δεν σας έχω γνωρίσει όλους, γι' αυτό θα συστηθώ. Είμαι ο Κλάους Χάινερ Λένε. Από το 2016 είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και επανεξελέγει για άλλα τρία χρόνια. Η θητεία μου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας 28 μέλη, τα οποία όλα ε, έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό και διαφορετικό ρόλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να συναντήσουμε κάθε ένα από εσάς ε, και ελπίζω να ε, μπορέσουμε να σας ε, ε, καλωσορίσουμε στο Λουξεμβούργο. Να δούμε λιγάκι τι με ενδιαφέρει σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί θέλω να σας παρουσιάσω την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ετήσια έκθεσή μας και κυρίως με την δήλωση αξιοπιστίας αξιολογούμε κατά πόσον τα κονδύλια τα οποία εσείς ως Κοινοβούλιο εγκρίνατε πέρυσι στον προπολογισμό, κατά πόσον τα κονδύλια αυτά δαπανή ε, με κάποια λογική και όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Ε, δηλαδή, πολύ σύντομα θα σας πω ότι είμαι λιγάκι σαν γιατρός, ε, θα κάνω μία αξιολόγηση και θα σας πω ποια τμήματα του οργανισμού λειτουργούν σωστά, πού ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα και πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα. Ο συνάδελφος κύριος Λάζαρος Λαζάρου είναι επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος έχει εξετάσει διάφορα στοιχεία των αιτήσεων λογαριασμών, τις δαπάνες και τα έσοδα. Ερεύνησαν αυτές, αυτούς τους υπολογισμούς και έτσι λοιπόν ε, κατέληξαν σε απόψεις για τον προεπλισμό του 2018. Αποκινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη καταλήξαμε με απόλυτη ειλικρίνεια στο τι ακριβώς ε, πρέπει να γίνει και τι ακριβώς έγινε. Μετά από τις ε, παρατηρήσεις σας, ε, φαντάζομαι ότι έχετε, κάνει, έχετε δημιουργήσει και εσείς μια εικόνα. Η αξιολόγησή μας αφορά όλες τις πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Όπως και κάθε χρόνο, και φέτος ε, ο ετήσιος ε, προϋπολογισμός ε, του 2018 εξετάστηκε από εμάς και ως εκ τούτου τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται ακριβώς όπως είναι, ικανοποιητικά, δεν παρουσιάζουμε καμία στρεβλή εικόνα. Με βάση τις παρατηρήσεις μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να υπολογίσει και να συμπεριλάβει και να ενισχύσει τις διαδικασίες που αφορούν συνταξιοδοτήσεις. Βεβαίως, όσον αφορά το συνταξιοτικό, θα συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Δεύτερον, Όσον αφορά στα έσοδα του ευρωπαϊκού προεπλογισμού, δεν διαπιστώσαμε σημαντικό ποσοστό λάθους ασχοληθήκαμε με το σύστημα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το σύστημα αυτό διασφαλίζεται ότι οι διάφορες πηγές εσόδων, οι πηγές αυτές υπολογίζονται σωστά και δηλώνονται σωστά. Εκτός αυτού εξετάσαμε και μία σειρά άλλων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εσόδων. Εξετάσαμε και εθνικά συστήματα. Επισκεφτήκαμε τρία κράτη, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Σε αυτές τις χώρες πήγαμε αυτή τη φορά και στις τρεις αυτές χώρες διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά στους δασμούς. Και επιπλέον διαπιστώσαμε ότι ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους, ο έλεγχος αυτός δεν βασίζεται ε, σε αξιολόγηση κινδύνου. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδείγματο χάρη ε, δεν προβαίνει σε αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο και δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσον οι έλεγχοι αφορούν κυρίως εκείνους τους τομείς όπου υπάρχουν οι περισσότεροι κίνδυνοι για τους ίδιους πόρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα έτσι ώστε να εκφράσει τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τα αποκαλούμενα στοιχεία BN Data η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μα, ε, διαπίστωσε ότι όσον αφορά κυρίω τη Γαλλία, στον τομέα αυτό υπήρχαν προβλήματα. Διαπιστώνουμε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρίτη κατά σειρά έτο έχει επιφυλάξει σε σχέση με του δασμού ε, που επέβαλαν τα, επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τι εισαγωγέ από την Κίνα. Τρίτον, όσον αφορά στο ποσοστό σφάλματο στι δαπάνε και αυτό αυτό βασικά διατρέχει το σύνολο της δήλωση αξιοπιστίας ε, και το 2018 αν διαπιστώσαμε το ποσοστό σφάλματος ανέρχεται σε 2,6%. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι 2,6% των πληρωμών ε, δεν έπρεπε να επιβαρύνουν τον ενωσιακό προϋπολογισμό γιατί οι ε, δαπάνες αυτές ε, δεν έλαβαν χώρα λαμβάνοντας υπόψη τους κείμενους κανονισμούς. Βεβαίως αυτή η αξιολόγηση συγκαλύπτει ένα βασικό γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι πληρωμές επηρεάζει πάρα πολύ τον κίνδυνο σφάλματος. Όσον αφορά τις δαπάνες οι οποίες υπόκεινται σε περίπλοκους κανονισμούς ε, που σημαίνει μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία και αυτό είναι κατ' ουσίαν το ίμιση του ενωσιακού προπολογισμού, έχουμε καταρχήν να κάνουμε με πληρωμές ε, που βασίζονται σε επιστροφές και τα αιτήματα για επιστροφή απορρέουν ε, ή γίνονται και ολοκληρώνονται με βάση και την ε, υποβολή δαπανών. Πρόκειται δηλαδή για προγράμματα τα οποία αφορούν την ε, γεωργική ανάπτυξη όπως επίσης και ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. Εκεί το ποσοστό σφάλματος ανέρχεται σε 4,4% κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Αντίθετα, ο κίνδυνος σφάλματος είναι χαμηλότερο ε, σε καταβολές που βασίζονται με βάση δικαιωματικές απαιτήσει. Εκεί η δικαιούχοι λαμβάνουν ένα ποσό αν καλύπτουν ορισμένες ε, προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη άμεσες καταβολές ε, σε γεωργούς, ε, υποτροφίες σε φοιτητέ ή χορήγηση βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Με άλλα λόγια, περίπου 50% των λογαριασμών που ελέγξαμε δεν παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό σφάλματος. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο για το τρίτο κατά σειρά έτος καταλήξαμε ε, σε ένα ναι, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις. Ε, θεωρούμε ότι είναι ενθαρρυντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κατά τα δύο προηγούμενα έτη ε, πράγματι σημείωσαν πρόοδο και επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν τομείς με πολύ λιγότερους ε, κινδύνους. Άρα δηλαδή ε, ο έλεγχος μας ε, ήταν τελικά θετικός. Παράλληλα βλέπουμε ότι υπάρχουν τομείς όπου εξακολουθούν να υφίστανται υψηλοί κίνδυνοι και αυτό μας ανησυχεί γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής πολιτούς στρατηγικής του, το ελεγκτικό συνέδριο προσπαθεί ε, την δήλωση αξιοπιστίας να την βασίσει και σε συγκεκριμένες δοκιμές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στο μέλλον θα εξετάσουμε τα ελεγκτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στα στοιχεία που τις δίνουν τα κράτη-μέλη. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν δρόμο ε, ικανοποιητικό, άρα δηλαδή καταρχήν να κάνουμε μετριοπαθή βήματα και αργότερα να επιδιώξουμε το στόχο να εκμεταλλευτούμε εργασία την οποία έχουν ήδη προσφέρει άλλοι. Από την ετήσια έκθεσή μας μπορείτε να διαβάσετε ότι πολλά από τα κράτη-μέλη, ε, πολλοί έλεγχοι που έγιναν από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ε, τους αντιμετωπίζουμε με κριτικό πνεύμα. Υπάρχουν 26 σημεία, τα οποία στον έλεγχο των δαπανών ε, συνοχής ε, συμμετέχουν σε αυτόν τον έλεγχο και αυτό πολύ συχνά μας δυσχεραίνει στο να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου και να μπορούμε να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα αξιόπιστα. Όμως θα ήθελα κατηγορηματικά να επισημάνω ότι οι ίδιοι ελεγκτές μας στο το σημαντικό τομέα της συνοχής έχουν διαπιστώσει και βελτιώσει για να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε την εργασία των ε, αρχών να μπορεί να την βελτιώσει περαιτέρω. Και ως εκ τούτου συνεργαζόμαστε, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να επιτύχουμε βελτίωση στους ε, ελέγχους και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Ότιγκερ και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που θα μπορέσω να συνεχίσω αυτή την εργασία με το διάδοχό του. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπής. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στη στις, στους διάφορους τομείς ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Όσον αφορά τον τομέα ανταγωνισμός, εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα σφάλματα από ό,τι πέρυσι. Έχουμε δαπάνες προσωπικού, εκεί εξακολουθούν να είναι τα περισσότερα σφάλματα. Επίσης διαπιστώνουμε ότι παρά τις ε, προσπάθειες ε, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να εξετάζει καλύτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί εκεί υπάρχουν τα περισσότερα σφάλματα ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο μία μικρομεσαία επιχείρηση που εφάρμοσε το πρώτο της project, ανέφερε δαπάνες 1,1 εκατομμύριο ευρώ, περίπου το 1 τρίτο ε, αυτών των δαπανών όμως ε, περιείχε σφάλματα και επίσης διαπιστώσαμε ότι ο έλεγχος όσον αφορά τις δαπάνες ε, μεγάλων δομών δεν μπορούσαμε να κάνουμε έλεγχο στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι παρότι υπήρχε παλαιότερα διεξοδικός έρευνος έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλα αυτά δαπάνες των 75.000 και των 30.000 ευρώ για μας ήταν αμφισβητή Όπω Όπως και πέρυσι σας καταθέσαμε μία γνωμοδότηση για ε, νομοθετική πρόταση. Εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να πλουστευτούν τα ερευνητικά προγράμματα. <clears throat> Κατά την άποψή μας, στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 μέχρι το 2027, στο πρόγραμμα Horizon, ορίζοντας, ε, κάποια ε, αίτια που οδηγούν σε σφάλματα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τώρα πλέον είναι καθήκον του νομοθέτη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίσουν πλέον αυτές τις νομοθετικές διατάξεις. Βεβαίως οι ελεγκτές μας είναι στη διάθεσή σας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά την ε, οικονομική και κοινωνική συνοχή, ένας άλλος ε, τομέας. Εκεί επίσης διαπιστώσαμε σφάλμα του 5%. Ε, τα λάθη που εντοπίσαμε καταδεικνύουν ότι όσον αφορά τις δαπάνες που παρουσίασαν τα κράτη-μέλη, οι δαπάνες αυτές εξακολουθούν να παρουσιάζουν αδύναμα σημεία. Έχουμε μη επιλέξιμες δαπάνες, αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και με τον τρόπο αυτό επιδεινώνεται το ότι διάφορα κράτη, εκτός από τις πολύπλοκες νοσιακέ διατάξει προσθέτουν και δικές τους διατάξει το περίφημο gold plating. Υπάρχει και ένα άλλος προβληματικό τομέα. Μία υπηρεσία μπορεί να αναθέσει χωρίς διαγωνισμό ε, ένα project και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα. Περίπου ένα σφάλμα της τάξης του 2,4% το οποίο αποτελείται από μη επιλέξιμες δαπάνες ε, στη γεωργία, ε, για ζώα, για εκτάσεις και αυτό συνδυάζεται και με άλλες μη επιλέξιμες δαπάνες. Αυτά Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν βέβαια και τομείς όπου δεν υπάρχουν μεγάλα σφάλματα. Είναι καλή αυτή η πληροφορία, αλλά τελικά ε, διαπιστώσαμε ότι μπορούν και να μειωθούν τα σφάλματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν καλά συστήματα ελέγχου. Οι γεωργοί θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους ε, online και ε, θα μπορούν να ελέγχονται online και τα στοιχεία που θα καταθέτουν. Αν πάμε όμως σε άλλες μορφές πληρωμής, διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις είναι πολύ πιο περίπλοκες και εκεί αυξάνεται ο κίνδυνος. Παραδείγματος χάρη, εξετάσαμε μία περίπτωση στην Πολωνία, όπου διάφορα μέλη της ίδιας οικογένειας κατέθεσαν ε, διαφορετικές αιτήσει για την κατασκευή ενός χειροστασίου ε, και ανέφεραν ότι πρόκειται για ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, εμείς διαπιστώσαμε ότι αυτή η οικογενειακή επιχείρηση τελικά δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση που κατά κανόνα χορηγείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στον τομέα της ασφάλειας, εκεί επισημαίνουμε αδυναμίες όσον αφορά τις διατάξεις ε, ε, ανάθεσης και ανάθεσης μετά από διαγωνισμό. Εδώ αναφέρομαι κυρίως τα ταμεία που υπάρχουν για την ασφάλεια. Αυτό ήταν ένα τομέα που ελέγξαμε. Εξ γνωρίζετε, στον τομέα Ευρώπη στον κόσμο προβλέπονται υψηλά κονδύλια και για μέλη ε, μέλη ε, ΜΚΟ. Αυτή τη φορά είχαμε προγράμματα τα οποία έγιναν από την UNICEF και από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής. Εκεί όμως υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν κατατέθηκαν έγκαιρα τα στοιχεία. Κατά τη δική μας άποψη αυτή η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα σε διεθνείς οργανισμούς όταν ε, πρόκειται για την υποβολή στοιχείων και εγγράφων εφόσον τα ζητούμε. Αυτό είναι απαράδεικτο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ευγνώμων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή ε, εγκρίνει τη σύστασή μας και για διεθνείς οργανισμούς προβλέπει ένα σύστημα της άμεσης λήψης επαφής. Οι ελεγκτές μας επίσης έλεγξαν μία σειρά περιπτώσεων μη επιλέξιμων δαπανών. Ε, Παραδείγματο χάρη ένας διεθνή οργανισμός ο οποίος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε 31 αεροπορικά εισιτήρια. Είναι προφανές ότι αυτό είναι μια επιλέξιμη δαπάνη. Τέλος, το ποσοστό σφάλματος για τον τομέα της διοίκησης και εκεί υπήρξαν αρκετά σφάλματα και θέλω να επισημάνω κυρίως δύο θέματα. Καταρχήν ελέγξαμε και είδαμε πολλές αδυναμίες όσον αφορά τον έλεγχο των οικογενειακών επιδομάτων προς τους ενωσιακούς υπαλλήλους. Ε, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Διαπιστώσαμε επίσης πολλά σφάλματα όσον αφορά τους ελέγχους που έκανε το Κοινοβούλιο για την ε, βελτίωση της ασφάλειας των κτηρίων μετά τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν συμφωνίες πλαίσιο που είχαν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με μία και μόνο προσφορά να μπορεί να ανατεθεί ένα έργο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με ένα μόνο ε, συμμετέχοντα σε διαγωνισμό. Ε, κατά την άποψή μας όμως ε, δεν υπήρχε πήγουσα κατάσταση για να ανατεθεί διαγωνισμός χωρίς άλλους ενδιαφερόμενους. Και ε, τελικά πέρασαν και πάρα πολλοί μήνες ε, χωρίς να δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Πριν ολοκληρώσω, θέλω να σε επισημάνω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεργασία με εσά. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής, ε, την οποία δρομολογήσαμε σήμερα το πρωί, είμαστε στη διάθεσή σας και εκτός αυτού είμαστε πρόθυμοι σε κάθε μία ειδική έκθεση που ενδεχομένως ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε. Η ε, κατατεθήσα έκθεση αφορά τα προηγούμενα έτη. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, έχουμε μία νέα θητεία, έχουμε ένα κράτος μέλος που πρόκειται να αποχωρήσει και τα υπόλοιπα 27 κράτη ε, συνεχίζουν τις ε, διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 21 έως 27. Ε, αυτά που σας παρουσίασα σήμερα το το πρωί, οι έλεγχοι για τους οποίους μίλησα καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, σφάλματα, για τρίτο κατά σειρά έτος η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι απόλυτα διαφανής όσον αφορά την χρήση κοντιλίων. Από τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε ότι θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες, ότι θα ε, προσπαθήσει να άρει τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ο κύριος Λαζάρου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή και σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ε, εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίδεται. Νομίζω ότι καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου ή θέλετε ε, να τον δώσω στον κύριο Ότιγκερ. Στον κύριο Λαζάρου. Όχι, τότε στον κύριο Ότιγκερ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Λένε, αξιότιμα μέλη της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε για όλα αυτά που μας είπε. Τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Τον ευχαριστούμε για τα συμπεράσματά του, ε, τα οποία και συμμεριζόμαστε. Είμαστε ευγνώμονες για το ότι κατά, για 12ο κατά σειρά έτος έχουμε ε, ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα οικονομικά μας σε γενικές γραμμές βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Το ποσοστό σφάλματος τα τελευταία χρόνια μειώθηκε σημαντικά. Το 2018 ε, μιλάμε για 2,6%. Ε, πριν από λίγα μόνο χρόνια μιλάγαμε για διπλάσιο ποσοστό σφάλματος και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το χαμηλό ποσοστό σφάλματος ε, να το τηρήσουμε ή αν θέλετε να μειώσουμε ακόμα περαιτέρω το ποσοστό αυτό. Για τρίτη κατά σειρά χρονιά το ελεγκτικό συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά το σύνολο των δαπανών δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα και αυτό είναι μια εξέλιξη που είναι πολύ σημαντική. Κατά τα άλλα ε, θα εξετάσουμε το αποτέλεσμα όλων των προγραμμάτων για να δείξουμε ότι υπάρχει υπεραξία ε, σημαντική αυτή για μας όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές επενδύσεις. Μιλάμε για εκατομμύρια που αφορούν ε, τους ερευνητές, τους νέους ανθρώπους, τους γεωργούς, ε, τους δήμους, τις κοινότητες. Για όλους αυτά τα οικονομικά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μία πολύ σημαντική σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι αυτή που λέει ότι όσον αφορά αυτά για τα οποία πρέπει να απολογηθούμε, εκεί ισχύει η αρχή και πρέπει να ισχύει η αρχή ένας και μόνο έλεγχος στα διαχειριστικά συστήματα. Και εισήχθη αυτή η αρχή. Δηλαδή, ακόμα και αν ε, τα κονδύλια δόθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές ε, από τις Βρυξέλλες, παρόλα αυτά υπάρχει μία και μόνο δομή, η ρόλη είναι σαφής... Ε, ε, είναι υποχρέωση να υπάρχει διεξοδικός έλεγχος. Ε, ένα ατού αλλά και μία δυναμία της Ευρώπης είναι η επικουρική μορφή διαχείρισης. Σε πάρα πολλά προγράμματα ε, δεν δραστηριοποιούνται οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα Υπουργεία, στα κράτη-μέλη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ή τα Δημαρχία ή αν θέλετε και άλλοι θεσμοί όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Ερυθρός Σταυρός ή οποιοδήποτε άλλος διεθνής οργανισμός. Αυτό είναι και αλλοι θεσμοι οπω ειναι η παγκοσμια τραπεζα ο ερυθρο σταυρο η οποιοδηποτε αλλο διεθνη οργανισμο αυτο ειναι και δυναμία. Το ατού είναι διότι επί τόπου έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία στι Βρυξέλλε, έχουμε μια εταιρική σχέση ανάμεσα σε δημόσια διοίκηση, εδώ δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη πλευρά το Προεδρείο, ε, ο εξειδικευμένος οργανισμός. Και από την άλλη πλευρά η αδυναμία είναι ότι εξαρτώμεθα από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα υπαλλήλων και συνεργατών άλλων υπηρεσιών, άλλων κυβερνήσεων. Ας πάρουμε το θέμα των ιδίων πόρων και ε, το τι σημαίνουν οι ίδιοι για τον ε, δικό μας ε, τον προπολογισμό. Ο κύριος Λένε έφυξε το θέμα της αξιολόγησης των κρατών μελών με βάση την ύπαρξη κινδύνου. Αυτό το θέμα θέλω να το δείτε λιγάκι πιο προσεκτικά. Για φανταστείτε, έχουμε 27 κράτη που τα αξιολογούμε τα εξαιρετικά, τα μέτρια, τα μη ικανοποιητικά, τα αρνητικά. Αν το κάναμε αυτό, τότε οι ευρωβουλευτές από τις χώρες που τα αξιολογούμε αρνητικά θα ερχόντουσαν σε εμά και θα λέγανε πώς τολμήσατε να το κάνετε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν να είστε σίγουρος ε, ότι εκεί όπου γνωρίζουμε ότι οι διοικήσει ε, δεν είναι αποτελεσματικές, είναι διεφθαρμένες ή έχουν διαφορετική ερμηνεία από ότι εμείς, όπως στο θέμα Ηνωμένων Ηνωμένο Βασίλειο και δασμοί, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, είμαστε πιο προσεκτικοί, εμφανιζόμαστε πιο συχνά, χωρίς όμως ε, να αποδίδουμε χαρακτηριστικά, γιατί νομίζω αν το κάναμε αυτό, τότε θα θέταμε σε κίνδυνο την ε, συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης είναι σαφές ε, ότι τα προγράμματα ενίσχυσης ε, από μόνα τους ενέχουν πολλούς κινδύνους. Έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις ε, με δημάρχους, με ευρωβουλευτές και σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζεται ένα θαυμάσιο πρόγραμμα το οποίο είναι επιλέξιμο. Για σκεφτείτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να θεωρηθεί μη επιλέξιμο. Όλοι λένε ότι είναι τα προγράμματά τους επιλέξιμα. Εγώ όμως είμαι πολύ πολύ επιφυλακτικός ε, και έναντι των ε, ευρωβουλευτών. Κατανοώ πολύ καλά ότι προσπαθούν να βοηθήσουν ε, το δήμαρχο της περιοχής τους, παραδείγματο χάρη, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα επιλέξιμα προγράμματα ενέχουν πάρα πολλού κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν το δικό μα το καθήκον είναι να χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια, αλλά επίση ε, οι οδηγίε ε, να είναι κρυστάλλινε ω προ τον ορισμό του. Ε, υπάρχει ένα θέμα για το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027. Αυτό το θέμα για μένα είναι η απλούστευση. Εγώ επιθυμώ οι κανόνες να απλούστευτούν στον ερευνητικό τομέα, παραδείγματος χάρη, γιατί εκεί πολλές ε, μικρές επιχειρήσεις ε, μας είπαν ότι ούτε καν κάνουν τον κόπο να ζητήσουν κονδύλια, γιατί είναι πολύ τεράστιος ο κόπος. Πρέπει λοιπόν να επιφέρουμε την απλούστευση και θέλω να παρακαλέσω το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις τομεακές προτάσεις να μην περιπλέξει τα πράγματα γιατί συνήθως οι ε, πρόταση Κομισιόν στο τέλος ήταν πολύ πιο περίπλοκη μετά από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου που συμπεριλαμβάνονταν όσο πιο πολύ απλουστεύουμε την κατάσταση ε, τόσο πιο εύκολο είναι δυνατόν να αποτρέψουμε ε, το ενδεχόμενο των καταχρήσεων. Όσον αφορά την αξιολόγησή μας των σφαλμάτων, βασιζόμαστε σε λεπτομέρειες, ε, ξεκινάμε από τη βάση, ε, πολλές λεπτομέρειες, κάνουμε και εμείς δικούς μας ελέγχους και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσο υψηλό είναι το ποσοστό των δαπανών που μπορεί να συμπεριλαμβάνει σφάλματα. Γνωρίζουμε ότι οι δαπάνες αυτές ε, θα μπορούσαν στο μέλλον να, μάλλον οι δαπάνε με σφάλματα θα μπορούσαν να είναι μικρότερες ε, εάν ε, καλούντο τα κρατημέλη να επιστρέψουν τα χρήματα. Δηλαδή το ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο και μετά από τον έλεγχο όλων και μετά από την διεξαγωγή όλων των ελέγχων το ποσοστό σφάλματος περιορίζεται και θεωρούμε ότι ε, στο τέλος αυτό που απομένει ως σφάλμα το 2018 είναι κάτω από το 1%. Είναι περίπου 0,8%. Χαιρετίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο από κοινού με εμάς ε, θα συμπεριλάβει όλα αυτά υπόψη του στη νέα δήλωση αξιοπιστίας. Όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, είμαστε όλο και πιο κοντά, συγκλίνουν οι απόψεις μας. Το ελεγκτικό συνέδριο πλέον ε, μπορεί να ελέγξει κατά πόσο μπορεί να βασιστεί στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία νέα δήλωση εξοπιστίας, μία νέα DAS, ε, τα ίδια κριτήρια, μπορεί να τα υιοθετήσει αν θέλει το ελεγκτικό συνέδριο και πάνω σε αυτά να προβεί στις δικές του, στα δικά του συμπεράσματα. Στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Εκεί συνεργαζόμαστε για να υπάρχει μια νέα προσέγγιση και σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής θα επεκταθούμε και εκεί. Όπως το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι και εμείς ε, για το 2018 ε, διαπιστώνουμε αυξημένο αριθμό προβλημάτων, κυρίως όσον αφορά στην πολιτική της συνοχής. Θα έλεγα ότι σχεδόν σε όλα τα άλλα προγράμματα το ποσοστό σφάλματος μειώνεται, αλλά στην πολιτική συνοχής πέρυσι εμφανίστηκαν νέα προβλήματα. Και ε, αυτό το βασίζουμε σε λεπτομερείς πληροφορίες, τις οποίες πήραμε από τη βάση. Έτσι λοιπόν, πέρυσι είχαμε συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση προγραμμάτων συνοχής σε αρκετά κράτη-μέλη. Συνολικά, ε, σε αρκετές δαπάνες συνοχής εμφανίζονται σφάλματα το ελεγκτικό συνέδριο επισήμανε κάποια θέματα. Συνεργαζόμαστε όμως με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο λόγος δεν είναι ότι δεν είναι καλοί οι υπάλληλοι που δουλεύουν επί τόπου, αλλά το ότι καθυστερούν στην εφαρμογή τους τα προγράμματα, ότι μόλις το 17 άρχισαν να εφαρμόζονται, το ότι για τις διοικήσεις τώρα πλέον υπάρχουν περισσότερα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν, να ελεγχθούν, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πολύ περισσότερα το 17 από ότι το 16 ή το 15. Και συμφωνούμε επίσης με το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπάρχουν ιδιαίτερα περίπλοκες διατάξεις που αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο του σφάλματος. Ένας ε, έλεγχος. Ένας έλεγχος δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο. Σε ορισμένα θέματα εμείς ε, έχουμε διαφορετική άποψη από ότι το ελεγκτικό συνέδριο και γι' αυτό λοιπόν σε πέντε περιπτώσεις, μόνο σε πέντε περιπτώσεις ε, δεν καταλήξαμε στην ίδια άποψη ε, την οποία έχουν και οι ελεγκτές του ελεγκτικού συνεδρίου. Είμαστε σε συνεχή διάλογο με το συνέδριο. Πρόκειται κατ' ουσίαν για το εξή πώς εν μέρη εθνικές διατάξεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για προγράμματα και για ενίσχυση, πώς πρέπει να ερμηνεύονται νομικά αυτές οι διατάξεις. Και εδώ πάλι βιώνουμε την πολυμορφία της Ευρώπης. Ε, έχουμε ε, ευρωπαϊκές ε, βάσεις, sectoral proposals, αλλά αυτές συμπληρώνονται εν μέρη με εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις. Ω εκ τούτου, η πολυμορφία εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. Ο κύριος Λίν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις. Αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εμείς θα τις ελέγξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι κατά πόσον τα διοικητικά και ελεγκτικά συστήματα, κατά πόσον αυτά ελέγχουν, έτσι ώστε τα σφάλματα να είναι μία μικρή εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Γι' αυτό και εμείς είμαστε ευγνώμονες για το ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει καταθέσει μία σειρά θετικών προτάσεων, παρήματος χάρη στον ε, γεωργικό τομέα, όπου επιτύχαμε πρόοδο και εκεί ε, κατά κανόνα η εφαρμογή είναι πολύ καλύτερη. Γενικά λοιπόν το ποσοστό σφάλματος ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι χαμηλό. Για τη τελική ανάλυση για τον φορολογούμενο εκείνο που μετράει είναι το ποσό το οποίο δόθηκε λανθασμένα και δεν μπορεί να ε, αναζητηθεί, να επιστραφεί. Μιλάμε για ένα 0,8%. Όσον αφορά την ε, απόδοση, για μας και για το Κοινοβούλιο η υπεραξία είναι πολύ σημαντική. Για μας ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις και εδώ βεβαίως δεχόμαστε τις προτάσεις της δικής σας Επιτροπής αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αυτήν την έκθεσή μας περί επιδόσεων δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει. Μπορούμε βεβαίως να βελτιωθούμε περαιτέρω όσον αφορά τι οικονομικέ μας επιδόσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι δείκτες ε, ε, δεν είναι οι καλύτεροι και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με διάφορους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε ε, να βελτιώσουμε περαιτέρω τους δείκτες στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πάντα με ένα κοινό στόχο δηλαδή ε, να παρουσιάσουμε στον ε, φορολογούμενο τις βέλτιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που πρέπει να απορρέουν από τον προπολογισμό και με τον τρόπο αυτό να παρουσιάζεται η βάση για σωστές πολιτικές. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Λένε, τον κύριο Λαζάρου, το ελεγκτικό συνέδριο στο σύνολό του. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας, ε, για τον τρόπο με τον οποίο μας συνδράμετε. Ε, θεωρώ ότι η συνεργασία αυτή είναι επικοδομητική. Η συνάδελφός μου και εγώ ε, και η επόμενη επιτροπή ε, θα προβούμε σε συγκεκριμένα βήματα. Είναι ημερομηνίε σαφείς. Ε, νομίζω θα δείτε κι εσείς ότι το 2018 μπορεί να παρουσιαστεί με πολύ καλή, με, χωρίς πρόβλημα στον Ευρωπαίο πολίτη το ε, Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχουν ένα και μόνο στόχο να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό σφάλματος και να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω ε, το θέμα των οικονομικών επιδόσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ότιγκερ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή, μάλλον να τους καλωσορίσω, τη Γενική Διεύθυνση Προεπολογισμών. Σας ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία των τελευταίων ετών, γιατί με τον τρόπο αυτό κατορθώσαμε να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος από 4,8% στο 2,6%. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε πάρα πολλούς τομείς επιτύχαμε ε, σημαντικά αποτελέσματα και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι ακολουθούμε έναν ικανοποιητικό δρόμο. Εγώ προσωπικά ως ε, εισηγήτρια θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μένα, στην υποφαινόμενη και στους ε, εισηγητές. Και να πω δύο πράγματα. Έχουμε ε, δύο θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Πρώτον, να δούμε κατά πόσον οι δαπάνες ήταν νομότυπες, κατά πόσον τηρήθηκαν οι διατάξεις ε, και κατά πόσον οι επιστροφές ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσον και αυτές ε, είναι νομότυπες, κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για τους στόχους για τους οποίους είχαν προβλεφτεί. Κατά τα άλλα, έχω να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. Διαπιστώνουμε ότι ε, το να υπάρχουν δύο διαφορετικές διοικήσεις ή διοικήσεις σε διάφορα επίπεδα, αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή τα προγράμματα δεν τα εξετάζει μόνο το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο κατ' ουσίαν ελέγχει το πώς ε, έλεγξαν οι εθνικές αρχές, αν ήταν σωστή η διαδικασία που ακολούθησαν, ε, εξετάζει δηλαδή, το ελεγκτικό συνέδριο τη δυνατότητα των κρατών μελών για διεξαγωγή ελέγχων. Ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου είπε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, ταξινομηθούν με βάση τους υφιστάμενους κινδύνους. Ο Επίτροπος βέβαια φοβήθηκε, τρόμαξε και είπε «επουδενή» ε, και θα ήθελα ως εκ τούτου να ερωτήσω μήπως ακριβώς επειδή ε, για τόσα πολλά χρόνια εξετάσαμε όλο το κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Μήπως γι' αυτό είχαμε υψηλό ποσοστό σφάλματο. Όχι ότι θέλω να πω ότι ένα κράτο μέλο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ω ιδιαίτερα επικίνδυνο, αλλά πράγματι υπάρχουν κάποιε εθνικέ αρχέ, ε, ε, οι οποίε ήταν καλύτερα από άλλε, λιγότερο έμπειρε. Βεβαίω ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Για μένα το να αξιολογήσουμε με βάση τον κίνδυνο αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ κάποιον, απλά ε, θέλω να πω ότι μπορεί να το δει κανεί και αλλιώς. Δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη διοίκηση δεν επωφελείται όσο θα μπορούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτά που υποβάλλει είναι συνδυασμένα ε, με ένα μεγάλο ποσοστό σφάλματος. Και τελικά, εμείς οι Ευρωβουλευτέ, ε, τι μας εξυπηρετεί αυτό, τίποτα. Μένουν χρήματα αδιάθετα ή δίδονται με λάθο τρόπο και ε, τελικά ο πολίτης δεν επωφελείται. Να σας υπενθυμίσω την περίπτωση της Σλοβακίας, η φαρπαγή γης, η Ρουμανία και εκεί υπάρχει το θέμα της φαρπαγής γης. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν στην Ουγγαρία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα και τους δύο και τις δύο πλευρές να τις ερωτήσω το εξής. Μήπως θα είχε νόημα να σκεφτούμε κάποια άλλα εργαλεία πέρα από αυτά που ήδη διαθέτουμε και ποια εργαλεία θα ήταν κατάλληλα όχι μόνο για να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος αλλά πράγματι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ενωσιακά κονδύλια. Ποια μέτρα κατά την αποψία πρέπει να ληφθούν. Κατόπιν, έχω και ένα ερώτημα σχετικά με τις 126 διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες ε, συμμετέχουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, στον έλεγχο. 126 είναι πάρα πολλές. Βέβαια, είναι και πολλά τα προγράμματα αλλά τελικά τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι 126 υπηρεσίες ε, είναι ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα αυτά. Συντονίζονται οι υπηρεσίες. Με ενδιαφέρει να ξέρω ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα. Κυρίως όσον αφορά, επαναλαμβάνω, στι 126 διαφορετικές υπηρεσίε. Κατόπιν, ποσοστό σφάλματο, Ο Επίτροπο και εγώ πριν από μερικέ ημέρε, είχαμε ανταλλαγή απόψεων ως προς το ότι εγώ κατανοώ ότι υπάρχει ποσοστό σφάλματος μετά τη διόρθωση, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι και το ποσοστό σφάλματος το οποίο καταλήγει το ελεγκτικό συνέδριο μετά την επιστροφή κονδυλίων. Άρα δηλαδή στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε δύο ποσοστά, διαφορετικά ποσοστά σφάλματος. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι αδυναμίες. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο πού καταλήγει, σε ποιο ποσοστό σφάλματος μετά την επιστροφή κονδυλίων. Γιατί από εκεί θα μπορούσαν να προκύψουν διαρθρωτικές αλλαγέ και να εξάγουμε και συμπεράσματα για το τι πρέπει να αλλάξει και στις εθνικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ανακαλύπτει η Κομισιόν και από τη μία πλευρά και το ελεγκτικό συνέδριο από την άλλη, το κενό αυτό, η διαφορά αυτή να σμικρινθεί. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει είναι όσον αφορά τις ε, συστηματικές αδυναμίες. Με ενδιαφέρει αυτό. Αυτές οι συστημικές ή συστηματικές αδυναμίες, ε, κατά ποιες ακριβώς είναι. Ε, όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, το ότι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί δεν υποβάλλουν σχεδόν ε, κανένα στοιχείο, αυτό εκνευρίζει πάρα πολύ, γιατί χρειαστήκαμε μήνες ολόκληρους για να πάρουμε κάποια στοιχεία από την UNRWA, ε, παραδείγματος χάρη και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πράγματι πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερες μεθόδους συνεργασίας με αυτούς τους ε, διεθνείς οργανισμούς, γιατί το Κοινοβούλιο όταν απειλήσει με περικοπή κονδυλίων, ξαφνικά έρχονται όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, που καταλήγουμε ότι τα στοιχεία υποβάλλονται μόνο αν ε, ασκηθεί πίεση. Συστηματικά, οι διεθνείς οργανισμοί δεν μας δίνουν στοιχεία και αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τη συνεργασία μας. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουν στοιχεία. Και το τελευταίο, ε, το οποίο με απασχολεί, είναι το εξής. Κατά την άποψή σας, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούμε να πιστοποιηθούμε, αν θέλετε, σε εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Madam. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν απαντήσω σε αυτά που θίξατε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ για τη συνεργασία και για την πολιτική του προσήλωση για να κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση για τη δήλωση αξιοπιστίας. Για τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενδεχομένως ε, δεν είναι πλήρως εξοικειωμένα με αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια. Να σας πω ότι στο παρελθόν για τους σκοπούς της συμμόρφωσης εμείς επιλέγαμε τυχαία τις δικές μας συναλλαγές και ακολουθούσαμε τα κονδύλια μέχρι τον τελικό δικαιούχο. Και έτσι είχαμε μια εικόνα της διαδικασίας, της κατάστασης συμμόρφωσης ε, για κάθε χρόνο. Τώρα με τη νέα αυτή ε, διαδικασία δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο έργο των εθνικών ελεγκτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς όμως να ε, ε, δυσκολεύουμε πολύ τα πράγματα για τους δικαιούχους. Δηλαδή κάνουμε μία αναθεώρηση κινδύνου ή ελέγχου και όπου αυτό είναι απαραίτητο επαναδιενεργούμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο Έτεγκερ για την πολιτική βούληση να κινηθούμε προς την πλήρη τέτοια διαδικασία ελέγχου και χαιρετίζουμε την βελτιωμένη συνεργασία και με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρησιακό επίπεδο για να πετύχουμε το σκοπό μας. Πράγματι υπάρχουν ζητήματα στον τομέα της συνοχής και ένας τρόπος να επιληθούν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη όταν θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όμως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει το σύστημα ελέγχου της. Το είπαμε λοιπόν στην ετήσια έκθεση ότι η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος κατά την πληρωμή είναι 1,7% από πλευράς Επιτροπής. Ποσοστό συγκρίσιμο με το δικό μας ποσοστό σφάλματος το 5%. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει το έργο της. Θα πρέπει να έχει στατιστικό δείγμα οριζοντίως και όχι απλώς να δέχεται ότι οι επενδύσεις χαμηλού κινδύνου έχουν μηδενικό σφάλμα. Γιατί ο τρόπο που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ποσοστό σφάλματο είναι ότι επικεντρώνεται στου κινδύνου, στου τομεί κινδύνου, βρίσκουν σφάλματα, δεν τα ανάγουν, δεν τα προβάλλουν στο ευρύτερο δείγμα και γι' αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με το δικό μα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Έτιγκερ και για αυτό που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Είμαστε πολύ σημαντικοί εταίροι. Και γι' αυτό, όπως και εσείς, και εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω της συνεργασίας. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να υπάρχει ακόμα περισσότερη συνεργασία συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ναι, μερικά σχόλια και από πλευρά μου για την ανάλυση κινδύνου στα κράτη-μέλη. Από πλευρά ε, εσόδων του υπερπολογισμού, ε, δεν έχω πρόβλημα με το πώς ε, κάνει τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκεί να ξέρει τι κάνει και βασίζεται στις ε, αρχές μας κάθε χρόνο. Αλλά έχουν ένα σύστημα που ε, πρέπει να έχουν ένα σύστημα το οποίο αναγνωρίζει και εντοπίζει τα προβλήματα και βοηθάει και την επίλυσή τους. Ωραία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε από πλευρά ε, ΦΠΑ, για παράδειγμα, εξετάζοντα την ανάλυση τη Europol, θα είχαμε ε, μεγαλύτερα επίπεδα ιδίων πόρων αν ε, παίρναμε τον ΦΠΑ όπως θα έπρεπε, αν τον εισπράταμε. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει και θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον να εντοπίσουμε πού ακριβώς υπάρχουν αυτά τα σφάλματα. Έχω κάποιες πληροφορίες από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που είχαν ε, ατέρμονες συζητήσεις και έρευνες. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στους Σκιώδης. Ματίνα Πάκοβα. Α, μάλιστα. Εδώ είστε δεν κοιτούσα στο σωστό σημείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ελέν και τον κύριο Λαζάρου που παρουσίασαν την ετήσια έκθεση. Ε, με ικανοποίηση ακούμε ότι ε, δίνεται ε, τέτοια θετική γνώμη για τις πληρωμές τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι θετικό που υπάρχει μείωση στα ποσοστά ασφάλματος για την ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και δεν υπάρχει αύξηση, δεν υπάρχει αύξηση στους φυσικούς πόρους. Ωστόσο, αυτοί οι δύο τομείς ακόμα παρουσιάζουν ουσιαστικό σφάλμα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα βελτίωσης. Ευχαριστώ κύριο Έτιγκερ για την παρουσία του εδώ και συμφωνώ απολύτως ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος είναι σχετικά χαμηλό και παρουσιάζει αρνητική τάση, μειούμενη τάση τα τελευταία χρόνια. Μετά υπάρχει το θέμα με τους ε, τομείς συνοχής που αναφέρεται πολύ σωστά. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει εντοπίσει σε δυναμίας, σε και κάποια ανησυχητικά δείγματα σε ορισμένε γενικέ διευθύνσει, όπω η Ριτζιο και η Άμπο. Και αναγνωρίσατε και τα ποσοστά σφάλματος ε, σε ό,τι αφορά του ε, τομεί κοινωνική συνοχή για το, τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2018 ω μία αξιόπιστα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το εξετάσουμε και να το βελτιώσουμε. Εσείς ποια μεγάλα προσκόμματα εντοπίζετε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προκειμένου να υλοποιήσουν την σύστασή σα για τη βελτίωση των ελέγχων, ιδίω στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, οι ασυνέπειε που έχετε εντοπίσει στις άμεσες ενισχύσει για την κοινή γεωργική πολιτική για το σχετικό ποσοστό σφάλματος. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν εκεί λέει ότι δεν εντοπίζονται σφάλματα στις άμεσες ενισχύσει. Όμως οι εκθέσει εκθέσεις της Γενικής Άγκρη εντοπίζει ένα σφάλμα 1,7%. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Και στρέφουμε και προς τους δύο εδώ. Και τέλος, Στο ψήφισμα για την απαλλαγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2017, το Κοινοβούλιο καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιοποιήσει τα αιτήσια προστασφάλματο για ε, την Global Europe και για την ασφάλεια. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε αυτή την έκθεση τώρα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζάρου. Ή ποιος θέλει να απαντήσει. Ναι, μάλιστα, να δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου. Ξεκινώ από το τελευταίο. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε μια στατιστική μέθοδο που σημαίνει ότι αντλούμε ένα δείγμα είναι σαν να κάνουμε μια δημοσκόπηση στην ουσία και να ρωτάμε τον κόσμο τι κόμμα θα ψηφίσει. Είναι αρκετά παρόμοιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα δείγμα συγκεκριμένου μεγέθου για να έχουμε στατιστικά σημαντική ε, απάντηση. Αν έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, τότε η στατιστική απάντηση δεν έχει κανένα νόημα. Αν ρωτήσουμε μόνο 38 άτομα τι κόμμα θα ψηφίσουν, δεν θα έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα. Πρέπει να ρωτήσουμε χίλια άτομα. Επομένω, αυτή η μέθοδο έχει αυτομάτω περιορισμού. Όπω και να έχει, ποτέ δεν μα φέρνει ένα ακριβέ νούμερο. Γι' αυτό μιλούμε για εκτιμόμενο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι πάντα υπάρχει ένα όριο μέσα σε αυτή την καμπύλη. Έχουμε 90% ε, πιθανότητα και συν πλήν 1%. Το πραγματικό ποσοστό σφάλματος είναι κάπου εκεί μέσα. Όσο είμαστε κάτω από ε, ένα συγκεκριμένο ποσοστό ε, σημαντικότητας, δεν δίνουμε τις πληροφορίες αυτές για το ποσοστό σφάλματος, γιατί ποτέ δεν είναι ακριβές. Είναι τόσο χαμηλό που δεν έχει νόημα να σας δίνουμε τέτοια στοιχεία. Εξαιτία τη στατιστική ε, μεθόδου, ποτέ δεν είναι ακριβή ο αριθμό, πάντα έχει ένα συγκεκριμένο όριο και στα παραρτήματα θα βρείτε τα στοιχεία. Αλλά στο βαθμό που μπορούμε να σας τα δώσουμε. Εκεί λοιπόν αν δείτε τα παραρτήματα θα βρείτε λογικά τα στοιχεία που θέλετε. Ότι είναι δηλαδή κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό μπορώ να σας πω προς το παρόν για αυτό το τεχνικό σκέλος. Μετά για τα εμπόδια και προσκόμματα να δώσω το λόγο στο Λάζαρο. Ναι, ποια είναι τα προσκόμματα, πώς μπορούμε να τα επιπηδήσουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, θέλουμε καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πάνω από 10 χρόνια συζητούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και το Κοινοβούλιο το λέει, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ελεγκτική προσέγγιση. Επιτέλους τα καταφέραμε και εμείς θέλουμε πραγματικά να την εφαρμόσουμε αυτή την ενιαία προσέγγιση. Λάβαμε μια στρατηγική απόφαση ότι θα πρέπει να κάνουμε και τις δικές μας, ε, τους δικούς μας ελέγχους ε, συναλλαγών, αλλά να αξιοποιούμε περισσότερο το έργο των ε, κρατών μελών και της Επιτροπής και θα επιμείνουμε σε αυτό. Ο Επίτροπος Έντιγκερ ανέφερε ότι είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πράγματι έτσι ξεκίνησε, αλλά θα παραμείνει, θα το διατηρήσουμε. Γιατί τα ποσοστά σφάλματος δεν είναι τόσο κοντά όσο είναι στην ανταγωνιστικότητα και στους φυσικούς πόρους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επιτυχία. Γιατί συλλέξαμε τις απαραίτητες ε, πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να δώσουμε, να παράσχουμε μία γνωμοδότηση ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα ε, φωτίζουμε αυτές τις αδυναμίες ε, του συστήματος ελέγχου που καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπεράσει. είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Για το τρίτο ζήτημα τώρα. Γιατί δεν σας παρουσιάζουμε ε, ποσοστό σφάλματος για την Global Europe, ε, την ασφάλεια και την ε, ευρωπαϊκή θαγένεια. Πράγματι, σημειώνουμε και λαμβάνουμε γνώση του περσινού αυτού ψηφίσματος απαλλαγής αλλά στην ουσία έχουμε πολύ περιορισμένους πόρους, τους οποίους θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από στατιστικής άποψης, λοιπόν, αποφασίζουμε πόσες συναλλαγές πρέπει να ελέγξουμε από τον ετήσιο προπολογισμό για να έχουμε 95% σιγουριά για τα στοιχεία που σας δίνουμε. Καταλήγουμε λοιπόν σε έναν ε, συνολικό αριθμό, τον οποίο διαιρούμε σε διάφο... και κατα... κατανέμουμε σε διάφορους ε, τομείς ε, του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Συνολικά οι τομείς που προανέφερα είναι 11 δις. Είναι πολύ χαμηλό το νούμερο για αυτούς τους τομείς λοιπόν για να κατευθύνουμε επιπλέον πόρους, επιπρόσθετους πέραν των πόρων που χρειάζονται για να έχουμε εικόνα συνολικά για τον προπολογισμό. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτούς τους πόρους μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα. Δεν έχει νόημα να δώσουμε δηλαδή ποστό για αυτούς τους ε, τομείς. Όμως, έχουμε ειδικέ εκθέσεις για αυτούς τους δύο τομείς. Δεν είναι σαν να τους ε, αμελούμε τελείως να παραγνωρίζουμε αυτές τις ε, δαπάνες. Δίνουν πληροφορίες μέσω των ειδικών εκθέσεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σούστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε της ετήσιας έκθεσης και επίσης να χαιρετήσω την εργασία που έχει κάνει το ελεκτικό συνέδριο στο σύνολό της. Η παρουσίαση που μας έγινε σήμερα ε, ξεκινά για μας την διαδικασία απαλλαγής. Βρισκόμαστε δηλαδή στην αρχή των συζητήσεων και των εργασιών μας. Αυτό που θέλω να κρατήσω από την πρώτη ανάγνωση ε, του θέματος είναι το εξής. Φυσικά δεν είναι απλό να βρει κανείς την σωστή ισορροπία σε έναν προϋπολογισμό που θέλει να είναι και ορθολογικός αλλά και φιλόδοξος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει υποσχέσεις και πρέπει να τις διατηρήσει, να τις κρατήσει. Αυτό είναι και το μήνυμα άλλωστε το οποίο είχατε δώσει και τον προηγούμενο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω την βούληση του ελεγκτικού συνεδρίου για περισσότερους ελέγχους ε, ε, μέσω των οποίων θα μπορέσει να ελεγχθεί το κατά πόσον εφαρμόζονται σωστά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά τους δείκτες επίδοσης. Κάθε ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και αποτελεσματικά, ε, γιατί εδώ παίζεται και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της και των θεσμών της. Και βεβαίως ε, θα θέλαμε στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία επίδοσης. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι απεδείχθη από τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ότι δεν υπάρχει πολύ ε, ε, μεγάλο ποσοστό ε, σφάλματος. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει και κάποιες επιφυλάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρξε το ίδιο επίπεδο αποτελέσματος σε όλα τα στοιχεία του ελέγχου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δειχθεί ιδιαίτερα προσοχή σε ορισμένα σημεία. Προβλήματα τα οποία δεν είναι καινούρια και όπου όμως από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρνουμε, αργούμε ε, να ε, ελέγξουμε. Όπως ας πούμε το θέμα των επιστροφών. Εκεί έχουμε ε, ποσοστό σφάλματος μεγάλο. Επίσης σε ορισμένες χώρες μικρό ποσοστό απορρόφησης. Αναφερθήκατε εσείς στο gold plating, αυτήν την επιβολή επιπλέον υποχρεώσεων. Επίσης οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από την Κομισιόν δημιουργούν κάποια προβλήματα. Ε, επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Ανάπτυξης, ε, όλα αυτά είναι προβλήματα, ενδεχομένως όχι πάρα πολύ μεγάλα, ωστόσο που επιμένουν επί σειρά ετών. Και αυτό καταδεικνύει ότι θα πρέπει να κάνει διορθωτικές πράξεις η Κομισιόν. Ερώτηση. Ποια μέθοδο θα πρέπει να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε ε, το ποσοστό λάθος εξειδικευμένα στις δαπάνες υψηλού κινδύνου. Πολύ σημαντικό. Επίσης, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες στατιστικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις απάτες. Υπάρχουν προγράμματα όπου στατιστικά ε, ε, διαπιστώνεται μεγαλύτερος αριθμός απατών. Τέλος, πώς εξηγείτε και ποιες είναι οι συμβουλές που μπορείτε να δώσετε όσον αφορά την, το μεγάλο ποσοστό σφάλματος ε, στις δαπάνες συνοχής έρευνας, καθώς επίσης και προγράμματα όπως είναι το Erasmus ή το ε, Horizon 20, 2020. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, απαντήστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαστέλ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει με αρκετά απλό τρόπο για, τον, για την πρώτη και τρίτη ερώτηση η συνοχή και έρευνα γιατί εκεί υπάρχουν ε, ζητήματα μα γιατί ε, πρέπει να πω ότι είναι περίπλοκη όλη η διαδικασία, όλη η διαδρομή είναι περίπλοκη. Και όσο πιο περίπλοκες είναι, ε, περίπλοκοι είναι οι κανόνες, τόσο πιο δύσκολη είναι η εφαρμογή. Ε, είπαμε προηγουμένως ότι 126 υπηρεσίες ε, πρέπει να ελέγξουν. Δεν λέω ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος, γιατί αριθμητικά, ποσοτικά η έλεγχη είναι πολύ. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερο έλεγχο. Όπως ε, το είπαμε άλλωστε και την προηγούμενη χρονιά, δεν χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι, αλλά καλύτερα ποιοτική έλεγχη, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θα πρέπει να ξαναδιαβάσω. Τι μας είπατε, ποια ήταν η δεύτερη ερώτησή σας. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορούσε τις ε, απάτες και τους τομείς ε, στους οποίους ε, το ποσοστό απάτης ήταν μεγαλύτερο. Ναι, ναι, ναι, το θυμήθηκα τώρα. Όσον αφορά τις απάτες, λοιπόν. Εμείς είδαμε εννέα περιπτώσεις, νέες περιπτώσεις και ε, ε, υποχρεωθήκαμε να έρθουμε σε επαφή με την Όλαφ γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες υποψίες απάτες. Η ΔΕ Όλαφ αποφάσισε να ελέγξει περαιτέρω δύο περιπτώσεις για τις υπόλοιπες ε, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας σύμφωνα με τις διαδικασίες Όλαφ. στις 728 ε, ε, διαδικασίες είχαμε μονάχα 7 ε, υποψίες απάτης. Ε, επομένως ε, το ποσοστό είναι μικρό για τόσο μεγάλο αριθμό συναλλαγών. Ε, επομένως, ε, κατά την άποψή μας ε, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Όμως, ίσως θα πρέπει να υποβάλλετε αυτό το ερώτημα στον Όλαφ, γιατί αυτή είναι η υπηρεσία που γνωρίζει καλύτερα τα θέματα της απάτης και είναι η υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να σας πει με τα βεβαιότητος ποιοι είναι οι τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά απάτης. Πάντως, για φέτος δεν μπορούμε να σας δώσουμε κάποιο άλλο μεγάλο αποτέλεσμα γιατί ήταν τρία της χιλής. Επομένως, πραγματικά κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Βιόλεφαν Κράμον ε, θα έπρεπε να υποβάλει την ερώτηση, αλλά η συνάδελφος αυτή λείπει. Ε, μήπως έχει δώσει κάποια στοιχεία. Ναι, ναι, θα πάρω το λόγο. Εξ ονοματός της. Πολλά υπόθηκαν ήδη από τους προελίσσαντες ε, συναδέλφους εισηγητές. Ίσως μια ερώτηση προς την ε, Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, είχαμε ε, μακρά συζήτηση για τα ποσοστά ασφάλματος και τα ασφάλματα γενικώ. Ε, η επεξήγηση η οποία δόθη και από το ελεγκτικό συνέδριο μου ακούγεται λογική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται αυτά. Θα ήταν πολύ περίπλοκο να υπάρξει μια διαδικασία αναφοράς, ένα reporting ε, ε, σχετικά με τα ποσοστά ασφάλματο ε, και στην έκθεση της Κομισιόν είναι υπερβολικά δύσκολο τεχνικά. Όμως, έχω και άλλη μία ερώτηση. Uh, Όσον αφορά το backlog, εάν καταλαβαίνω καλά, Υπάρχει ένα 36% αύξηση όσον αφορά ε, την ε, ε, δέσμευση των ποσοστών κονδυλίων υποχρεώσεων σε σχέση με το 2011. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά χρήματα ακόμα τα οποία θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί στο παρελθόν και που περιμένουμε να καλυφθούν είτε από τωρινές ε, τωρινά έσοδα είτε από μελλοντικά. Ε, αυξάνεται όμως αυτό το ποσοστό, αυτά τα ποσά και επομένως ε, ελοχεύει συστημικός κίνδυνος να ξεμείνουμε κατά κάποιο τρόπο από ρευστό. Εγώ με προβληματισμό διαβάζω στη σελίδα 16 της σύντομης έκθεσης ε, πόσο αυτές ε, οι πιστώσεις υποχρεώσεων αφορούν την κάθε μία χώρα και το ποσοστό της 100, μάλλον ποια είναι η σχέση μεταξύ των πιστώσεων υποχρεώσεων και του συνολικού προϋπολογισμού των κρατών μελών. Ας πούμε για την Κροατία είναι 23%, για τη Βουλγαρία επίσης και 20% ε, για τη Λιθουανία, τη Λετωνία, 17% για την Πολωνία. Είναι πολύ αρκετά υψηλά ποσοστά αυτά. Εάν ε, κατάλαβα καλά, σε περίπτωση που ξεμείνουμε ας πούμε από ε, ρευστό, τότε θα υπάρξει πρόβλημα στις χώρες. Πρόβλημα αντίστοιχο ε, με αυτό που αντιμετωπίσαμε με την ε, δημοσιονομική κρίση του 2009. Μου φαίνεται μάλλον επικίνδυνο αυτό. Και ε, καταδεικνύεται αυτός ο συστημικός κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτόν τον κίνδυνο όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η πορεία αυτή με τον ίδιο τρόπο που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό ή πώς αντιμετωπίσετε κάποια κρίση αν και αυτή προκύψει. Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα απ' όλα να απαντήσει ο Επίτροπος ε, κύριος ε, και μετά θα δώσω το λόγο και σε άλλους και οδησηγητές. Όσον αφορά στο πώς ακριβώς ε, παρακολουθούμε και αντιμετωπίζουμε τα κράτη-μέλη που κάνουν λογιστικούς ελέγχους, να σας πω το εξής, ότι οι δικοί μου συνεργάτες βρίσκονται παντού εκεί όπου με βάση ενδείξεις ε, καταλήγουμε στο ότι μπορεί να έχει γίνει ε, κάποιο λάθος όσον αφορά τις καθαρίσεις των προγραμμάτων. Το θέμα της παροχή συμβουλών. Αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πολύ συχνά κάνουμε τέτοιου είδου ε, συναντήσεις, ακόμα και όταν προετοιμάζονται τομεακές προτάσεις, έτσι ώστε ή δυνατόν ε, να ε, βελτιώσουμε το επίπεδο για το πώς ακριβώς πρέπει να εφαρμόζονται οι έλεγχοι. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, το ποσοστό σφάλματος δεν σημαίνει απάτη δεν σημαίνει απαραίτητα δόλο. Ε, κατά κανόνα δεν υπάρχει δόλος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διαφοροποιούμε ανάμεσα στις περιπτώσεις των οποίων επιλαμβάνεται η Όλαφ και των άλλων ε, περιπτώσεων όπου εμείς ή το λεκτικό συνέδριο ενημερώνουμε την Όλαφ και η Όλαφ πλέον αποφασίζει πώς ακριβώς ε, θα αντιμετωπίσει αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, με το ενδεχόμενο της απάτης ή της ε, απιστίας. Του χρόνου μην ξεχνάτε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεσολαβεί και αυτή, θα παίζει και αυτή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως λοιπόν αναφέρθηκε πολύ σωστά, αυτό που τώρα έχει καθοριστική σημασία είναι η απλούστευση και εκεί είσαστε συνεργάτες μας. Εμείς προσπαθούσαμε να, προσπαθήσαμε να πλουστεύσουμε τους κανόνες, γιατί είναι σαφές ότι όσο πιο απλή είναι οι κανόνες, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ε, Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι διευκολύνεται η απάτη, που σημαίνει ότι ένας απλός κανόνας οδηγεί σε εφαρμογή χωρίς λάθη, αλλά ε, θα μπορούσε πράγματι να αυξηθεί και ο κίνδυνος απάτης, ε, γιατί ορισμένοι περίπλοκοι κανόνες ε, βασίζονται στο ότι υπήρχε πρόθεση εκ των προτέρων να μην υπάρχει δυνατότητα απάτης. Αλλά αυτό που σας λέω τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι το Κοινοβούλιο και ε, το ελεγκτικό συνέδριο στις 44 δικές μας προτάσεις να μην προκύψει επικάλυψη, το περίφημο gold plating, ε, και τα κράτη-μέλη να μην πρέπει απαραίτητα να προσθέτουν εθνικές ή περιφερειακές προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ε, άμεσες πληρωμές ε, προς τους γεωργούς, ένας γεωργός που έχει δύο συνεργάτες, 40 εκτάρια και 40 γελάδες, αυτός ειλικρινά εκνευρίζεται πάρα πολύ όταν έχει να κάνει ε, λογιστικά βιβλία, να τηρήσει λογιστικά βιβλία, να ελέγξει στοιχεία, να κάνει ελέγχους και αυτό να το κάνει κάθε χρόνο. Και γι' αυτό όσο πιο πολύ έχουμε πρασίνισμα και βιώσιμους στόχους, τόσο πιο πολύ θα έχουμε και συνεργάτη τον Γεωργό. Ε, στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει για το πώ ακριβώ το θέμα τη γεωργική πολιτική και οι ε, άμεσε ενισχύσει ε, προ του γεωργού, η κλιματική αλλαγή, πω όλα αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε σε ένα πλαίσιο που να είναι αποδεκτό για το γεωργό. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τη συνεργασία με τους ε, διεθνείς οργανισμούς ε, στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε θεσπίσει ικανοποιητικούς κανόνες που πρέπει να τηρήσουμε. Κανόνες βέβαια τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν και οι εταίροι μας. Ε, έγινε λόγος για περαιτέρω στοιχεία. Κοιτάξτε, εμείς ό,τι θέλετε μπορούμε να σας το παρέχουμε και εάν αυτή η Επιτροπή πει ότι για το 2018 θέλουμε και άλλα στοιχεία, προφανώς και θα σας τα δώσουμε. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο τεκμηριωμένο όσο το κάνουμε εμείς. Στα περισσότερα κοινοβούλια οι εθνικοί βουλευτές θα εκπλησόντουσαν εάν παίρνανε αυτό το έγγραφο που σας δείχνω. Εγώ στο Βερολίνο, στο, στη Στουτγάρδη, ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε καλοί, καλύτεροι από άλλους, μπορούμε βέβαια να βελτιωθούμε, αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και προσωπικό. Να μην ε, ε, βάζουμε κι εμείς στον εαυτό μας υπερβολικές απαιτήσει, γιατί αν θέλετε και άλλα στοιχεία, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει και άλλος χρόνος εργασίας, περισσότερες απαιτήσει έναντι των κρατών μελών, περισσότερη διοίκηση. Ε, ας μην το παρακάνουμε, ας προσπαθήσουμε να βρούμε μία μέση οδό. Αναφέρθηκαν ε, τα αδιάθετα ποσά, τα ραλ. Αυτό ε, είναι ένα θέμα που αφορά όλους ε, κάθε χρόνο. Τα υπόλοιπα προσεκαθάριση, τα ραλ, εμείς τα τεκμηριώνουμε. Βεβαίω ε, στον ε, προπολογισμό αναφέρονται οι πληρωμέ. Αν πλήρωσε κάποιος ε, το 16 κάποιο ποσό, δεν σημαίνει ότι μετά θα πληρώσει κάτι λιγότερο. Έχουμε τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές οι οποίες έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της συνοχής. Έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται και κάθε υπουργό γνωρίζει τι πρέπει να μας καταβάλει τα επόμενα πτέτη. Δεν γνωρίζει ακριβώς πότε. Ίσως ε, αυτό να πρέπει να γίνει το 20 το 22, αλλά όποιος ε, έχει καλό προϋπολογισμό γνωρίζει ότι μπορεί να πάρει από εμά κάποια ανταλλάγματα και ε, μπορεί να πάρει κάποια στοιχεία μόλις μας καταθέσει τα στοιχεία. Το πρόβλημα είναι ότι στην πολιτική συνοχή τα προγράμματα καθυστερούν και κάποια στιγμή έρχονται οι λογαριασμοί. Για το 2015 δεν πήραμε τόσους πολλούς λογαριασμούς. Τώρα παίρνουμε πολλοί περισσότερους. Το πρόβλημα του 12, 13, 14, εκεί ε, ήταν πολύ λιγότερα τα στοιχεία και καλούμε τα κρατη να μας υποβάλουν στοιχεία. Αλλά για άλλη μια φορά σας λέω, όλα αυτά για το φορολογόμενο δεν γίνονται ακριβότερα. Τα 7 χρόνια δεν υπάρχουν ε, εκπλήξεις. Τα 7 χρόνια, για 7 χρόνια καθορίζονται ήδη τώρα ε, τα στοιχεία μόνο δεν ξέρουμε ποια ακριβώ ημερολογιακή χρονιά θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε. Το τελευταίο, όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη γεωργία, το 1,8% αφορά το σύνολο των γεωργικών προγραμμάτων και τον, ε, ε, τον ε, δεύτερο πυλώνα. Το 0% αφορά τις άμεσες πληρωμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τελευταίο ηγητής, ο κύριο ε, Κούς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ελένε. ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ έχω μόνο μία παρατήρηση να κάνω και δύο ερωτήσεις. Η παρατήρησή μου είναι η εξή. Αυτό το 0,8% το οποίο ανέφερε ο κύριος Επίτροπος ε, ως ε, χρήματα τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν. Πρόκειται για προγράμματα που κάπου πήγαν στραβά και όπου δεν μπορούν να ανακτηθούν κονδύλια. Μιλάμε για ένα 0,8%. Αυτό ηχεί πάρα πολύ καλό, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 0,8% αντιστοιχεί σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ως εκ τούτου αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Έχουμε κονδύλια ε, τα οποία ε, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας επισημάνω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας έτσι ώστε να μην έχουμε ένα 0,8% που δεν μπορούν να ανακτηθούν, αυτό να πάει σε 0%. Ξέρω ότι το παλεύετε και θα ήθελα και εγώ να βοηθήσω. Ε, δύο ερωτήσεις. Μία λεπτομέρεια, δεν το κατάλαβα καλά, ε, αφορά την έκθεσή σας, ε, την, το ευσύνοπτο αυτό έγγραφο που διανύματε, συγκεκριμένα σελίδα υπαριθμών 7, κάτω από την επικεφαλίδα που λέει «Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός του 2018 ο νοσιακός προπολογισμός, στην τελευταία πρόταση, δεύτερη παράγραφος, γίνεται λόγος για 2,2% του συνόλου των δαπανών του κράτος ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ε, ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της την χαρακτηρίζεται ως ένα και μόνο κράτος. Ίσως μπορείτε λιγάκι να μου το εξηγήσετε. Αυτό ήταν μια ερώτηση κατανόησης. Δεν ξέρω, ίσως να είναι και λάθος ε, μετάφραση. Ε, Σα παρακαλώ πολύ να κάνετε ερωτήσει που να αφορούν τη δική μας Επιτροπή, την ΚΟΝΤ, όχι γενικέ ερωτήσει. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά ε, ένα μεγάλο πρόβλημα το πώς ακριβώς ε, καταλήγεται στο αποτέλεσμα των ε, δειγματοληπτικών ελέγχων. Μας μιλήσατε για δειγματοληπτικούς ελέγχους, ε, πώς κατόπιν κάνετε τις αναγωγές και καταλήγετε σε κάποιο συμπέρασμα. Άρα δηλαδή το συμπέρασμα δεν είναι το απόλυτο, αλλά είναι μία πρόβλεψη κατά προσέγγιση πρόβλεψη ε, παρόλα αυτά ε, καταλήγεται σε έναν ε, αριθμό, σε ένα στοιχείο το οποίο από το οποίο συμπεραίνει κανείς ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά όμως όλα που μας λέτε ε, θα πρέπει να είναι μία ενότητα. Και με όλα αυτά τα ε, διαφορετικά στοιχεία, τα διαφορετικά προγράμματα, ε, δικαιούχους, οργανισμούς, νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα νέο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, πώς μπορείτε εσείς να έχετε ένα δειγματοληπτικό, ένα δείγμα το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό για το σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τσιντόφσκι ε, θέλει να πάει σε μια ψηφοφορία, γι' αυτό του δίνω τώρα το λόγο. Συγγνώμη συνάδελφο, εφόσον ε, έχουμε τον ε, κύριο ε, στην άλλη αίθουσα, έρχεται σύντομα η σειρά μου να πάρω το λόγο, πρέπει να φύγω λοιπόν σύντομα. Ευχαριστώ όμως πολύ, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που ο Επίτροπος ε, πολλές φορές δείχνει τη βούληση να μας μιλήσει. Ανοιχτά και για τη διαδικασία ελέγχου. Πρώτο ερώτημα προς εσάς, κύριε Λένε. Το θέμα της συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Όλαφ. Ξέρω ότι πολλές φορές έχετε συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία ε, στο πλαίσιο του ΕΑΖΟ. Μπορείτε να μας πείτε για το μέλλον πώς θέλετε να ενισχύσετε αυτή τη συνεργασία. Δεύτερον, προς τον ε, Επίτροπο Έτιγκερ περισσότερο. Πρέπει να δούμε το ποσοστό σφάλματος και το σύστημα που χρησιμοποιείτε εσείς και υπάρχει διαφορετικό σύστημα το συνέδριο σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος. Στο μέλλον θέλετε να έχετε το ίδιο ελεγκτικό σύστημα. Ξέρω ότι δεν είναι πρόβλημα μεθοδολογίας. Αλλά και πάλι, αν το ελεγκτικό συνέδριο έχει 20% ποσοστό σφάλματος και εσύ έχετε μόνο 5-10%, υπάρχει πρόβλημα, γιατί κάτι υπολογίζεται ως φάλμα και κάτι άλλο όχι. Τρίτο ζήτημα για τη διαφάνεια. Εν γέννη υπάρχουν ε, προβλήματα με κάποια προγράμματα στην ε, πολιτική συνοχής, ιδίως ό,τι φορά τον ε, γεωργικό τομέα. Είδαμε αυτό το πρόβλημα και στη Σλοβακία και σε πολλά άλλα κρατημέλη. Εσείς τι θέλετε να βελτιώσετε στο μέλλον για να ενισχύσετε τους ελέγχους και να αποτρέψουμε έτσι τα σφάλματα σε κάποια κρατημέλη. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Τις απαντήσεις θα τις ακούσω μέσω της εφαρμογής στο κινητό μου. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Ich gebe sofort weiter an den Präsidenten. Gut, ich fange an und gebe dann einfach... Λοιπόν, ε, ξεκινάω και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου. Ε, κοιτάξτε, δεν έχω μπροστά μου τη γερμανική εκδοχή, αλλά έχω την αγγλική και εκεί λέει το 2,2% του συνόλου των κυβερνητικών δαπανών των κρατών μελών. Κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ότι ε, πρόκειται για τις δαπάνες ε, στο σύνολο των δαπανών σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το 2,2% το δίνουμε στο δημόσιο, ε, έτσι αναφέρεται και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του ΑΕΠ λοιπόν και γι' αυτό δεν μιλάμε για ένα κράτος, αλλά μιλάμε για τις ε, δαπάνες, δημόσιες δαπάνες όλων των ε, κρατικών δομών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από την εθνικότητα. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά ε, τη στατιστική μέθοδο, που όλες έχουν αδυναμίες. Αν δει λοιπόν κανείς τις μεμονωμένες συναλλαγές, αναγκαστικά θα δούμε και αυτό νομίζω ο Στάνφος κ. Λαζάρου το είπε, ε, στο με 95% πιθανότητες μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το πραγματικό ποσοστό σφάλματος ε, πλησιάζει περίπου το συν 1 πλην 1% του μέσου όρου. Γιατί υπάρχουν αυτές ε, οι καμπύλες τις οποίες έχουν επεξεργαστεί οι μαθηματικοί και το ποσό είναι στη μέση. Υπάρχει μια πιθανότητα κατά 95% 0,8 συν πλήν 0,8% να ισχύει η πρόβλεψή μας. Το 95% λέει ότι ε, το 5% ε, δεν ισχύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε διαφορετικά. Απλά πρέπει να κάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, μελέτες και αυτό απαιτεί περίπου το 40% των ε, πόρων μας. Άρα δηλαδή κάπου υπάρχει ένα όριο. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές ε, που λένε ότι κατά κανόνα μπορούμε να βασιστούμε ε, σε μια υπόθεση του 95%. Όλες λοιπόν οι στατιστικές μέθοδοι έχουν λάθη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού, αλλά δεν υπάρχει κανένα καλύτερο εργαλείο με, το οποίο, με το οποίο να μπορούμε να εργαστούμε. Άρα δηλαδή ε, κατ' ουσίαν δουλεύουμε με τις ε, ίδιες προδιαγραφές. Ε, ξέρω ότι δεν σας ικανοποιεί απόλυτα, αλλά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το σύστημα έχει πάρα πολλά λάθη, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όσον αφορά τις, ε, τα βασικά στοιχεία. Έχουμε τους ε, μαθηματικούς μας, οι οποίοι μας βοηθούν στη δημιουργία των προϋποθέσεων. Εγώ προσωπικά δεν είμαι μαθηματικός, είμαι νομικός, αλλά ε, νιώθω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι όλα γίνονται με επιστημονικά κριτήρια. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, ε, σχετικά με την ε, συνεργασία με την ε, Όλαφ, την, το άλλο σκέλος θα το απαντήσει ο κ. Λαζάρο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Όλαφ, έχουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο επεκτείνει τη συνεργασία και θα ήθελα να πω ότι ο νέος διευθυντής της Όλαφ ε, είναι ένα πρώην μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε και πολύ καλή προσωπική σχέση, υπάρχει χημεία μεταξύ μας, άρα συνεργαζόμαστε. Και θα προσπαθήσουμε, εφόσον ε, το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ε, θα συσταθεί και θα επαντρωθεί, θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με εκείνους αλλά βεβαίως είμαστε στην αρχική φάση. Υπήρξε η πρώτη ανταλλαγή επιστολών, όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν γιατί όλα αυτά είναι καινούργια και πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνεργασία. Αυτά είχα να σας πω και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Λαζάρου να απαντήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζενεχόφσκι για τις ερωτήσεις Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα υπολογισμού σφαλμάτων, δύο διαφορετικά μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καθορίζεται το σφάλμα ως τέτοιο εάν δεν ακολουθούνται οι κανόνες ε, και οι κανονισμοί. Ε, είναι παρόμοιο το ζήτημα. Μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Κομισιόν είναι αυστηρότερη στον προσυπολογισμό των σφαλμάτων, ας πούμε όταν μιλάμε για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Εμείς ε, είμαστε πολύ πιο επίοικείς ε, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης σε σχέση με αυτόν που έχει η Κομισιόν. Αυτό που, ε, στο οποίο ευθυγραμμιζόμαστε και πρέπει να ευθυγραμμιστούμε περισσότερο έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη δουλειά είναι, για παράδειγμα, ε, η, ε, ο έλεγχος των συναλλαγών επί στατιστικής βάσεως έτσι ώστε να υπάρχει αναγωγή. Γιατί η Κομισιόν δεν κάνει τέτοιου είδους ε, δοκιμές όπως το ανέφερα και προηγουμένως και δειγματοληψίες. Γι' αυτό λοιπόν ή μάλλον αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους εμφανίζεται αυτή η διαφορά κυρίως όσον αφορά τη συνοχή. Για την επόμενη ερώτηση τώρα, σχετικά με το πώς μπορούμε να προλάβουμε να αποτρέψουμε τα λάθη μέσω απλούστευσης μέσω ε, ε, ενισχυμένου, βελτιωμένου συστήματος ελέγχου και με ένα τρίτο τρόπο να μην προσθέτουμε ε, επιπρόσθετες υποχρεώσεις όπως ας πούμε για τις ε, πληρωμές της ε, γεωργίας έχουμε βάλει τώρα και κάποιες οικολογικές προϋποθέσεις και όπως είπε και ο Επίτροπος Ότιγκες προηγουμένως είναι πολύ δύσκολο για μια οικογενειακή επιχείρηση για έναν απλό γεωργό να υποβάλει όλα αυτά τα έγγραφα και να ακολουθήσει όλα τα βήματα τα οποία προκύπτουν λόγω των μέτρων αυτών. Επομένως, απλούστευση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο σε τρεις ερωτώντες, να είσαστε λίγο σύντομοι. Έχουμε ένα σκιώδη που επανήλθε, ο κύριος Τσανέτσκι, ε, Μούνιος και Λαμπαγιώβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη για δύο πράγματα. Πρώτον, ε, απουσίασα για λίγο, γιατί έπρεπε να ψηφίσω στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Και Ε, επειδή ακόμα δεν είμαι δυσυπόστατος, δεν μπόρεσα να είμαι και εδώ. Συγχαίρω τον πρόεδρο Λένε και τον κύριο Λαζάρου, γιατί πραγματικά ε, μας μίλησαν με τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χαίρομαι και χαίρομαι ε, γιατί έχει την Προεδρία ο κ. Λένε. Ε, όσον αφορά τις ε, εκτιμήσεις και τις αξιολογήσεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό και όσον αφορά τους, τους φυσικούς πόρους. Ακούσαμε αυτά που μας είπατε. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές και διαστάσεις όσον αφορά την ε, συνοχή. Διαπιστώνουμε δε ότι υπάρχει μια πτωτική ε, τάση όσον αφορά την συνοχή. ε, τουλάχιστον ε, το διαπιστώνουμε αυτό ότι για τον ε, νέο προπολογισμό του 20 έτσι θα είναι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Ε, αυτή είναι η γενική μου εκτίμηση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί μας είπατε και να μην ε, μακρηγορήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλετε να κάνω την ερώτηση τώρα. Ωραία. Ωραία. Θα προσπαθήσω να υποβάλω την ερώτηση που είχε Σκιώδης ε, για, τις ε, άλλες, ε, για τα άλλα θεσμικά όργανα. Και θα ήθελα μετά να κάνω και κάποια σχόλια. τα άλλα όργανα αναφέρονται στο κεφάλαιο διοίκηση και φαίνεται να υπάρχουν κάποια να μην υπάρχουν κάποια προβλήματα και δεν αναφέρονται και σημαντικά ποσοστά ασφάλματος. Επίσης, το κεφάλαιο ε, διοίκησης ε, αναφέρεται στο 9,9% του πιδελταπή και μονάχα το 2,1 αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα. Επομένως είναι πολύ μικρό το ποσοστό ε, και επομένως είναι κάτω από είναι πολύ μικρό ο κίνδυνος ε, και ακούσαμε και προηγουμένως, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν υπάρχουν πολλοί πόροι, ωστόσο ε, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έγιναν τόσο ε, μικρά δείγματα και μάλιστα βλέπουμε ότι τα δείγματα μειούνται από έτος προς έτος και επομένως ε, καταλαβαίνουμε βεβαίως αυτό που μας λέτε ότι το ποσοστό σφάλματος είναι μικρό αλλά ωστόσο αυξάνεται Ε, ε, έχουμε αύξηση γιατί από τις, το 2017 από τις 100 ε, περιπτώσεις είχαμε 12 ασφάλματα, το 2018 από τις 45 13 σφάλματα. Επομένως από το 12% έχουμε αυξηθεί, έχουμε ανεβεί πολύ περισσότερο. Τα παραρτήματα επίσης θα πρέπει να μελετηθούν σωστά γιατί νομίζω ότι και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για διαφάνεια και για διόρθωση της της ε, διοίκησης ε, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιολογούν βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ματίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ιδιαίτερα δεξοδική η έκθεση που αποδεικνύει και πάλι ότι παραμένει το ελεγκτικό συνέδριο ένας ε, ισχυρός και αμερόληπτος κριτής της, ε, των, της διαχείρισης των οικονομικών και των προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Εγώ πάντα είμαι υπέρμαχος ε, της ε, χρηστής διαχείρισης. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις επιδόσεις. Ε, συμφωνούμε με το κεφάλαιο 3 για το επόμενο πι δελτα πι θα πρέπει να γίνεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα προς το ελληνικό συνέδριο. Στην ετήσια έκθεση του 2017 το ελληνικό συνέδριο είχε διακρίνει ε, το ποστό σφάλματος ε, στις πληρωμές και στις ε, αποζημιώσεις, οι επιστροφές. Όπου το ποστό σφάλματος ήταν μόνο 2%. Στην ετήσια έκθεση του 2018 τώρα σημείωσε ότι αντί για το entitlement in the reimbursement, η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου χρησιμοποιεί τον όρο πληρωμές χαμηλού ρίσκου και πληρωμές υψηλού ρίσκου. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο όρων. Και δεύτερο ερώτημα και προς την Επιτροπή και προς το Δυτικό Συνέδριο. Κάθε χρόνο φαίνεται τα σφάλματα να είναι τα ίδια. Ε, μη επιλέξιμες προσωπικές δαπάνες, έμεσες δαπάνες, σφάλματα της εξαιτία του κανονιστικού υπερθυματισμού. Με όλη την κατάρτιση, τις κατευθυντήριες γραμμές, τη μεθοδολογία, την ανταλλαγή των πρακτικών και ούτε καθεξής. Πώς γίνεται μόνο το ελληνικό συνέδριο να εντοπίζει σφάλματα και όχι οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη ούτε στην Επιτροπή. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε μία και μόνο ελεγκτική διαδικασία από το ελεγκτικό συνέδριο και μόνο πριν την πληρωμή από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζάρου, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Γκαρθία Σαεμούνιοθ για τις ερωτήσεις. Πράγματι λοιπόν στο παρελθόν ελέγχαμε μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών. Στην πορεία όμως, καθώς προχωρούσαμε στον έλεγχο, τον προγραμματισμό μάλλον των ελέγχων μας, αποφασίσαμε να βασιστούμε στην πείρα που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα και στα αποτελέσματα των περασμένων ετών. Εδώ και αρκετά χρόνια λοιπόν αποφασίστηκε το ποσοστό σφάλματος στη διοίκηση ότι είναι μάλλον κάτω από το 2%. Κάτω από το ποσοστό σημαντικότητας. Τώρα αν είναι 1,8 είναι 0,6 δεν μας αφορά γιατί είναι κάτω από το όριο σημαντικότητας. Δεν αλλάζει κάτι. Προκειμένου λοιπόν να έχουμε την βέλτιστη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, είμαστε κάτω, λίγο κάτω από τις 50 συναλλαγές το χρόνο το οποίο είναι το στατιστικό δείγμα που χρειαζόμαστε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, προκειμένου να εκδώσουμε συγκεκριμένη εκτίμηση για αυτό τον τομέα του ΠΔΠ. Δεν είναι ελεγκτική γνώμη, είναι μία ένδειξη της κατάστασης ε, στη διοίκηση. Περνώ στο επόμενο ερώτημα. Πράγματι, ευσταθεί αυτό το ερώτημα που θέσατε. Η αλλαγή μεταξύ των δύο όρων από τα δικαιώματα και τις επιστροφές πήγαμε στα υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει διαφορά. Όπως ε, ανέφερα και προηγουμένως, κάνουμε τον προγραμματισμό μας βάσει των αποτελεσμάτων προηγουμένων ετών. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες υψηλού κινδύνου ουσιαστικά ε, ισοδυναμούν με τις επιστροφές, με τις δαπάνες επιστροφών. Υπάρχει και ένα μικρό τμήμα των δαπανών δικαιωμάτων που είναι υψηλού κινδύνου, παρότι τώρα μπορεί να μπαίνουν σε διαφορετική κατηγορία και το αντίστροφο. Η φετινή όμως περιγραφή, η τελευταία, είναι και η ορθή βάση των ε, στοιχείων που αποκομίσαμε τα προηγούμενα χρόνια από τους ελέγχους. Αν θα πρέπει να υπάρχει τώρα ένας και μόνο έλεγχος, μόνο από το Ελληνικό Συνέδριο, που να ελέγχει τις συναλλαγές, ε, τις εκθέσεις κτλ. Ναι, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει ενιαία διαδικασία ελέγχου. Γι' αυτό και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται στενότερα μαζί μας προς αυτό το σκοπό. Αλλά τώρα αν μπορεί τώρα το ελεκτικό συνέδριο να το κάνει μόνο του, αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε στα χωράφια της ε, ε, εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είμαστε ο ανεξάρτητος αμερόλητος ελεγκτής. Μήπως ο Επίτροπος θέλει να πει κάτι από αυτού. Κοιτάξτε, ε, βεβαίως έχουμε περιπτώσεις ε, που επανέρχονται και που περιλαμβάνουν σφάλματα. Θα μπορεί κανείς να διευθυνθεί Γιατί επαναλαμβάνονται τα σφάλματα. Διότι το ένα σφάλμα, παραδείγματο χάρη, ήταν το 17, ας πούμε, σε ένα ερευνητικό οργανισμό στο Γκράτς. Ε, το άλλο σφάλμα διαπιστώθηκε σε ένα άλλο Ινστιτούτο στο Ντέλφτ και το άλλο σε ένα Ινστιτούτο στο Μόναχο. Άρα δηλαδή έχουμε εκατοντάδες συνεργάτες οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτοί λοιπόν όλοι που υποβάλλουν ε, τις ε, αιτήσει τους ε, είναι αυτοί που κάνουν τα σφάλματα. Οι λιγότεροι κάνουν επαναλαμβανόμενα σφάλματα, αλλά κάνουν παρεμφερή σφάλματα κάποιοι άλλοι που έγιναν από κάποιους τρίτους. Άρα δηλαδή η παροχή συμβουλών βοηθάει. Ε, βοηθάει το να δίνονται συμβουλές ε, και από τα κράτη-μέλη στις περιφέρειες, παραδείγματος χάρη. Ε, θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ είπα στα πανεπιστήμια στην Βάδη Βίτεμβέργη πριν από κάθε αίτηση να συζητάμε έτσι ώστε να μην υποβάλλονται αιτήσει ε, από βοηθούς, αιτήσει ε, που έχουν λάθει και που τα ξέρει ένας ειδικό. Αλλά σας λέω, τα, ο ίδιος ο ετών ε, δεν υποβάλλει συχνά τα ίδια λάθη. Τα λάθη γίνονται από άλλους, τα σφάλματα δηλαδή. στο θέμα, παραδείγματος χάνει της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Αυτό είναι ένα νέο πρόγραμμα ναι, και σε ΜΚΟ και εκεί ισχύει αυτό που σας λέω, ε, δηλαδή ε, μπορεί να υπάρχει ένας ισπανικός οργανισμός προστασίας της φύσης που δεν ξέρει τίποτα από υποβολή αιτήσεων. Γιατί σας λέω, είναι εκατοντάδες ε, οι αιτούντες ε, και γι' αυτό είναι και πάρα πολλά τα ασφάλματα. Αν θέλει ε, το ελληνικό συνέδριο να κάνει αυτή τη δουλειά, πολύ ευχαρίστως. Θα πάμε και εμείς διακοπές. Μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν πάρουμε ένα πρόγραμμα στην στην Πάφο ε, και πρέπει κανείς να πάει από το Λουξεμβούργο στην ε, Λάρνακα ε, και μετά και δύο με το λεωφορείο, ε, καλύτερα να γίνεται ο έλεγχος από τη Λευκοσία. Άρα δηλαδή εξαρτώμεθα από τις, τους μικρούς δήμους και τις κοινότητες. Αυτή η αποκεντρωμένη δομή δουλεύει καλύτερα. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει ένα καθήκον να μας ελέγχει επικοδομητικά, αλλά και να μας παρέχει και συμβουλές. Ε, βέβαια, όχι στο εκτελεστικό, στον εκτελεστικό βραχίωνα. Εκεί σημασία έχουν οι περιφέρειες, οι Δήμοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί νομίζω ότι αυτή η δομή είναι πολύ αποτελεσματική. Βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Και κάτι τελευταίο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ε, στον τομέα 5, στην διοίκηση, εκεί έχουμε το 6% των δαπανών, όχι το 9,6, 6%. Και όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία και περιλαμβάνονται όλοι οι θεσμοί, όλοι τα κτίρια και οι συνεργάτες. Και στους συνεργάτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίζει τον κεντρικό ρόλο. Γι' αυτό εκεί έχουμε περισσότερες δαπάνες προσωπικού από τις ε, άλλους θεσμούς. Μιλάμε για ένα 6%. Ε, πολύ σωστό αυτό που είπατε. Προηγουμένως έγινε λόγος για 1,6. Μπερδεύτηκε αυτό το ποσοστό με το ποσοστό περί δαπανών. Λοιπόν, η Ματίνα έχει το λόγο και μετά η Αγγελική. Συγγνώμη, Επίτροπε, για τα σφάλματα. Αυτό που ρώτησα είναι πώς γίνεται μόνο το ελεγκτικό συνέδριο να εντοπίζουν αυτά τα σφάλματα και όχι οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατομελών. Και αυτό που είπατε είναι λίγο περάξενο, γιατί αν τα γνωρίζετε αυτά τα σφάλματα και ότι επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, γιατί δεν τα εντοπίζετε πριν το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ε, νομίζω αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι ξέρετε το λέω εγώ γιατί το έχω διαβάσει. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει κάποιους ε, τομείς ε, ρίσκου και ε, αν κάτι γίνεται εκτός αυτών των τομέων τότε προκύπτουν επιπρόσθετοι κίνδυνοι. Και το δεύτερο είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, στο πλαίσιο της, ε, του συστήματος εξετάζει και άλλους κινδύνους. Άρα δηλαδή ε, σε κάθε έλεγχο προκύπτει κάποια διαφορά. Εμένα θα με εξέπλητε να συμπίπτουν κατά 100% γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνεται στον έλεγχο. Αν προκύψει 0,0% απόκληση, εγώ θα έλεγα εδώ κάτι δεν πάει καλά. Θα υποψιαζόμουν ότι κάπου τα έχουν συμφωνήσει, τα έχουν βρει ή κάτι παρεμφερές. Ίσως ε, η συνάδελφος Μπίντσικ να λάβει το λόγο και στο τέλος η κυρία Βόλτερς. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όταν ένας πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαπιστώνει ότι ε, ένας οργανισμός ε, έχει κάνει κακή χρήση των κονδυλίων, τι γίνεται, πού πρέπει να στραφεί. Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση πραγματικά θα ταράξει τα νερά και θα συνταράξει μάλλον τους ε, Βρετανούς φορολογουμένους εξαιτία των δημοσιονομικών προεκτάσεων. Το ελεγκτικό συνέδριο με την έκθεση του βλέπει ότι το επίπεδο των ε, παρατυπιών έχει αυξηθεί το 2017, όχι μειωθεί. Και παρότι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο προπολογισμό έχει λάβει ε, γνώμη με επιφυλάξεις, όπως και να έχει, είναι θέμα σημαντικού προβληματισμού. Μόλις χθε έλαβαμε την έκθεση και εγώ πραγματικά ε, έχω, διατηρώ επιφυλάξεις ότι αφορά την ποιότητά της γιατί σε πολλά σημεία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει γνώμη. Για την Global Europe, λοιπόν, βλέπουμε ότι 9,5 δις έχουν ταπανηθεί σε πάνω από 100 χώρες και ούτε καν έχετε διατυπώσει γνώμη. Το ίδιο ισχύει για τα δημόσια οικονομικά των ε, χωρών εταίρων. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο δεν μπορεί να δώσει γνώμη για τα 885 εκατομμύρια βοήθειας σε τρίτες χώρε. Θεωρείτε ότι αυτό επαρκεί. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την πολιτικοποίηση του ελεγκτικού συνεδρίου, συνεχώς βλέπουμε ότι μπαίνουν πολιτικοί σε αυτούς τους ρόλους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σόφρον. Η έκθεση υπογραμμίζει και πάλι γιατί πρέπει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκάθαρα χωρί συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλουμε να πετύχουμε εγώ και το κόμμα του Brexit. Ε, από ό,τι φαίνεται ο καθένας ακολουθεί τους ε, δαίμονές του, πράγμα το οποίο βέβαια είναι λιγάκι προβληματικό. Ίσως, ε, συνάλφε Χεβερ, θα έχετε ακούσει ότι συγκεντρώνουμε ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις η κυρία Βόλτερς και μετά και οι τρεις ερωτήσεις θα απαντηθούν. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, για μια στιγμή στα ΡΑΛ, στα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Γιατί μεγάλο κομμάτι αυτών, νομίζω φέτος ήταν 280 δις που είναι τέτοια υπόλοιπα προ εκαθάριση, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν τα διεκδίκησε κανεί και ουσιαστικά πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία για του Ευρωπαίου πολίτε. Το ανέφερε προηγουμένω εν συντομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλούσαμε λίγο για τον κίνδυνο, κατά, πόσο υπάρχει ρίσκο για τον προπολογισμό. Όμω, εγώ θα σταθώ περισσότερο στο κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί προβληματικό αυτό το ποσό των 280 δι. Εάν το θεωρούμε λοιπόν μη ευκταίο αυτό το ποσό. Τι βήματα μπορούμε να πάρουμε για να μειώσουμε τα ραλ. Και κατά πόσο και από το ελληνικό συνέδριο υπάρχουν προτάσεις ε, και λύσεις. Πρόεδρος, Θέλετε να, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσετε πρώτος. Ναι, ναι. Κυρία Πίνσεφ. Όταν διαπιστώνει κάποιος ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Εάν πρόκειται για απάτη, φυσικά η ε, ποινικέ αρχές ε, μπορούν ε, να δραχθούν του ζητήματος και να αναλάβουν την εκαθαρίσή του. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο λαμβάνουμε ενδείξεις οι οποίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όχι φυσιολογικές. Και εμείς ανάλογα με την περίπτωση μεταφέρουμε τα θέματα στην Κομισιόν στην Όλαφ. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Ιβ, αυτό είναι πολιτική δήλωση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Όμως να πω το εξής, ε, βεβαίως κάθε κεφάλαιο μπορεί και πρέπει να ελέγχεται ε, υπάρχουν πολλές πληροφορίες και πολλές λεπτομέρειες, άρα θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ε, και μάλιστα σημαντικά. Ε, κάνοντας στατιστικές μελέτες έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε πόρους, ανθρώπινους, υλικούς κλπ. Δεν έχουμε τον προϋπολογισμό σαν ελεκτικό συνέδριο, έναν προϋπολογισμό χωρίς όρια. Άρα εμείς δίνουμε τις πληροφορίες που είμαστε σε θέση να συλλέξουμε και να δώσουμε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σωστά τις πληροφορίες. Και αν δούμε λίγο το παρελθόν, ε, θα διαπιστώσουμε τι γινόταν πριν από 20-25 χρόνια. Ε, έχουμε επιτύχει πολλά και για τρίτη ε, συνεχόμενη φορά μπορούμε να δώσουμε αυτήν την δήλωση αξιοπιστίας, τη βεβαίωση αξιοπιστίας χωρίς πρόβλημα. Ο κύριος Λαζάρου. Ο κύριος Λαζάρου παρακαλώ. Και μετά θα απαντήσει και ο Επίτροπος Σέτιγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χιβερέ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς ε, ως ελεγκτές βάσει της συνθήκης οφείλουμε να ε, ε, κάνουμε έναν έλεγχο επί του συνόλου και αυτό κάνουμε. Εάν επιλέξουμε συναλλαγές ή μάλλον όταν επιλέγουμε συναλλαγές από όλα τα πιδέλτα πι, αυτές ξεπερνούν το κατόφλι το οποίο έχει οριστεί και πρέπει να προκύψει ε, συγκεκριμένη ανάλυση για ποσοστό λάθους στο συγκεκριμένο πεδίο, το κάνουμε αλλά διαφορετικά επιλέγονται 150-160 ε, συναλλαγές ε, για ε, να ελεγχθεί το ποσοστό σφάλματος. Αυτό δεν είναι επιπλέον έλεγχος, αυτό δεν είναι στατιστικός έλεγχος, είναι επιπλέον έλεγχος. Είχαμε επίσης σε 728 συναλλαγές 64 υπό το κεφάλαιο Global Europe. Για να δώσουμε ποσοστό σφάλματος σε αυτό το πεδίο θα έπρεπε να αυξήσουμε τον αριθμό των συναλλαγών. Μακάρι να το κάναμε. Θα το κάναμε χωρίς πρόβλημα και να δώσουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ό,τι θέλει. Ωστόσο θα έπρεπε για να το κάνουμε αυτό ε, επιπλέον 200 ε, ε, εργαζόμενους και επομένως νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιούσαμε αν κάναμε κάτι τέτοιο σωστά τα χρήματα των πολιτών. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι εμείς καλούμαστε να δώσουμε έναν συνολικό έλεγχο επί του συνόλου Ε, τώρα, όσον αφορά την πολιτικοποίηση, κοιτάξτε, εγώ είμαι τεχνοκράτης. Εγώ μάλιστα είχα δουλέψει και στο Εθνικό Σύστημα Λογαριασμών στο, ε, στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έχω μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ελεγκτικό συνέδριο βασίζεται και εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα ε, λογιστικών μελετών, ε, καθώς επίσης εφαρμόζει και την δέουσα δεοντολογία. Ναι, έχουμε και κάποιους πολιτικούς μεταξύ μας, δεν το αρνούμε αυτό. We are a court, we are a college of 28 and we have a staff of about 900. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε, τι να σας πω, 900 ανθρώπους προσωπικό ε, που είναι πραγματικοί ε, auditors, επαγγελματίες ελεγκτές και οι οποίοι μελετούν και διερευνούν και κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του αποφάσεις, ούτε καν ο πρόεδρος δεν έχει τέτοια εξουσία. Εμείς ως κολέγιο αποφασίζουμε συνολικά. Κοιτάξτε, εγώ ε, είμαι επαγγελματίας, auditor, ε, Είμαι υπεύθυνος για την ετήσια έκθεση, ωστόσο δεν μπορώ να πάρω καμία απόφαση μόνος μου. Εγώ ε, στον τομέα μου θα πρέπει να αναφερθώ στα ζητήματα που έχουν προκύψει και μετά στην Ολομέλεια ε, που συνεδριάζουμε οι 28 ε, αναφέρω τα ζητήματα και θα προσπαθήσω να πείσω τους συναδέλφους για την ορθότητα των απόψεών μου και επομένως να έχω την, ε, το δικό τους πράσινο φως. Δεν είμαστε πολιτικοί και δεν εφαρμόζουμε πολιτικές αρχές στη διάρκεια του auditing. Λοιπόν, θα κάνω και εγώ ένα αστιακή ε, και θα πω ότι η πολιτική δεν είναι γεννημένη. Η πολιτική καλούνται να αποδείξουν ε, τι είναι με τη δουλειά τους. Και θα έλεγα και στο συνάλφα από την Αγγλία να διαβάσει την έκθεση του Βρετανικού Ελεκτικού Συνεδρίου. Ε, στην τελευταία έκθεση αναφέρεται ακριβώς το ποιες θα είναι οι συνέπειες της αποχώρησης ε, χωρίς συμφωνία. Στο ίντερνετ αναφέρονται 25 περιπτώσεις, δηλαδή συνέπειες για τα φάρμακα, στα φάρμακα, στα οικονομικά. Ε, δίδονται πολλές ε, συμβουλές στη Βρετανική κυβέρνηση. Ο μόνος ο οποίος μπορούσε να λάβει μία απόφαση ήταν ο κύριος Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποφάσισε να κλείσει το κοινοβούλιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ε, ούτε ο πρόεδρος Επιτροπής, ούτε το ελεγκτικό συνέδριο. Από ό,τι βλέπετε, η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά ε, στην Ευρώπη. Ε, φαντάζομαι μου επιτρέπετε να κάνω και κάποια αστιάκια. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Επίτροπο. Απευθυνόμενοι στον Βρετανό συνάδελφο, λέει η Πρόεδρος ότι πιο εύκολα μιλάτε από το να ακούτε αυτά που σας λένε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα των ραλ. Είναι ένα δομικό θέμα. Τρεις φορές το χρόνο ε, κατατίθεται μία έκθεση και εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τα λογιστικά, τους λογιστικούς υπολογισμούς των κρατών μελών. Ε, γίνεται αίτηση για ένα project, ανατίθεται το πρόγραμμα αυτό και μετά στο τέλος ακολουθεί η εκαθάριση. Και μόνο όταν έχουμε την εκαθάριση έχουμε και τη δυνατότητα με πληρωμές ε, να ικανοποιήσουμε τις ε, υποσχέσεις. Και λέμε στα κράτη-μέλη, παρακαλώ, να μην καθυστερείτε στις εκαθαρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί τα επόμενα τρία χρόνια οι πιστώσει πληρωμών είναι υψηλότερε από ό,τι τα προηγούμενα τρία χρόνια. Κυρίως όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη το Connecting Europe, ο, αερίου, χρειάζονται πολλές φορές μέχρι και έξι χρόνια. Υπάρχουν και καθυστερήσεις. Έχουν αναλυφθεί οι πιστώσεις υποχρώσεων, οι πραγματικέ πληρωμέ ακολουθούν αργότερα. Ο στόχο μα είναι βέβαια να υπάρχει κάποιο περιορισμό. Δεύτερον, για μένα είναι σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη ε, να δίδει τις πληροφορίε για κάθε ευρώ. Ε, κατά τα άλλα, θέλω να πω και το εξή. αν στις 19 Οκτωβρίου ο δικός σας ο ζητήσει παράταση, τότε θα είσαστε εδώ και θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις ε, στους επιτρόπους γιατί ε, οι επιτροποί έχουν ήδη οριστεί και θα ήταν πάρα πολύ καλό να μείνετε ένα χρόνο γιατί εκεί θα μπορούσατε να ρωτήσετε τους επιτρόπους οτιδήποτε θέλετε για αυτά που σας απασχολούν. Πρόεδρος, ο συνάδελφος φαίνεται ότι δεν τον νοιάζουν όλες αυτές οι πληροφορίες, δεν, δεν τον ενδιαφέρουν. Ε, σας ευχαριστώ θερμά και νομίζω ότι με αυτά τα πολύ χαριτωμένα που ακούσαμε μπορούμε νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα και πάμε στην, ε, στο σημείο υπαριθμών 4. Im Tagesordnungspunkt 4. Im Tagesordnungspunkt 4 äh, ε, στο σημείο υπαριθμών 4 ε, θα εξετάσουμε την περιπτωσιολογία ECA σχετικά με τη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Πίτροπο και τον Πρόεδρο του ηλεκτρικού Συνεδρίου. Der Sonderbericht des Rechnungshofes darf ich alle Beteiligten, die gerne reden wollen, nach αν έχετε τη ε, καλοσύνη, ε, μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα, γιατί δημιουργείται πρόβλημα στους υπόλοιπους συναδέλφους. Και εσείς κύριε Επίτροπε, και εσείς ε, αν έχετε την καλοσύνη και τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, σας ευχαριστούμε πολύ. θα ήθελα παρακαλώ και στην αίθουσα να κάνετε ησυχία ή δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συγγήτριά μας για αυτή την ειδική έκθεση είναι η κυρία Λάρα Βόλτας ε, και θα ήθελα όσον αφορά αυτή την ειδική έκθεση να δώσω το λόγο στην Εύα Λούντστρομ. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ που μου δίνετε το λόγο για να παρουσιάσω αυτή την ε, προσπάθεια για την βιωσιμότητα. Από το Συνεδρίου. Ονομάζομαι Εύα Λίνστρομ και είμαι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου από την 1η Μαρτίου του 2018. Μόλις ακούσατε την ετήσια έκθεση, όμως ε, είναι το ίμιση του έργου που διενεργείται στο Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί κάνουμε και ε, ελέγχους επιδόσεων και αναθεωρήσεις. Επομένως, εδώ θα σας μιλήσω για την ε, βιωσιμότητα και τις απαραίτητε ε, εκθέσεις. Να σας παρουσιάσω αρχικά το υπόβαθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κινητήριος μοχλός για το θεματολόγιο του 2030. Είναι λοιπόν εύλογο το να κοιτάξουμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Έχει κάνει πολλά το ελεγκτικό ε, συνέδριο στους τομείς του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, όμω είναι η πρώτη φορά που ε, εξετάζουμε ευρύτερα το θέμα των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το θεματολόγιο του 2030. Αφετηρία μας ήταν στην ουσία διτή ήταν αυτή η αφετηρία, αρχικά το θεματολόγιο 2030 βεβαίω. Έχουμε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με ένα ευρύ φάσμα στόχων, κλίμα, μεταφορές, καινοτομία και είναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι μόνο για τους υπολείπους, ε, τις χώρες που είναι μακριά από εδώ, ούτε μόνο για το κλίμα, αλλά για μια ε, ευρεία κλίμακα τομέων και σίγουρα αφορά και την Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν ε, δεσμευτεί να υλοποιήσουν ε, τους στόχους αυτούς και πολλά κρατημέλη υποβάλλουν εκθέσεις ε, για την πρόοδο που σημειώνουν. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν καλέσει την Επιτροπή ε, να πραγματοποιήσει μια τέτοια έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 μέχρι το 2019. Αυτή ήταν η αφετηρία μα λοιπόν αφενό. Αφετέρου, έχουμε την οδηγία. Βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, λοιπόν, κάποιε μεγάλε επιχειρήσει θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσει για τη βιωσιμότητα και το 2018 ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε υποχρέωση δημοσίευση. Σήμερα έχουμε 7.400 χώρε εισηγμένε στο χρηματιστήριο που πρέπει να υποβάλουν τέτοιε εκθέσει και η υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα δεν είναι κάτι το καινούριο στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια εξέλιξη που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί υπάρχει ζήτηση από πλευρά επενδυτών. Θέλουν να ξέρουν του κινδύνου βιωσιμότητα σε διάφορε εταιρείε και πώ ε, τη διαχείριση την χάνουν. Γιατί η κίνδυνη βιωσιμότητα είναι και κίνδυνη οικονομική. Αυτή η οδηγία έχει υλοποιηθεί με διαφορετικού τρόπου ε, στα επιμέρου κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, έχουμε αύξηση των, του αριθμού των ε, οργανισμών που έχουν υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Όμω, όλοι οι οργανισμοί πρέπει να βάλουν εκθέσει για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Φυσικά η δημοσιοποίηση έχει να κάνει με τη διαφάνεια Πρέπει κανείς να λέει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις και με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για τον ρόλο της ε, αξιοπιστίας. Γιατί φυσικά υπάρχει ένα οικολογικό προσωπείο παντού γύρω μας το βλέπουμε, αλλά είναι σημαντικό να είναι αξιόπιστες ε, αυτές τις πληροφορίες. Η οδηγία αφήνει ανοιχτό στα κράτη-μέλη τον ρόλο των ελεγκτών. Και λέει η οδηγία ότι οι ελεγκτές θα πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον ότι υπάρχει έκθεση βιωσιμότητα, χωρίς όμως να μπαίνει στο περιεχόμενο. Από αυτό το σημείο κίνηση, λοιπόν, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνει το σωστό παράδειγμα και να υποβάλει εκθέσεις για τις επιδόσεις της. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε ενωσιακό επίπεδο. Και πώς διενεργείται η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από επιμέρους ε, θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλούμε για το ενωσιακό επίπεδο σημαίνει ότι εξετάσαμε τον ενωσιακό προπολογισμό, όχι τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη, ούτε εξετάζονται εδώ μεμονωμένα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για αναθεώρηση, όχι για έλεγχο. Είναι μια τεχνική διάκριση. Αλλά στη δική μας επισκόπηση έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν το review να περιγράψουμε λοιπόν ε, την κατάσταση και να εντοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον. Εξετάσαμε λοιπόν τις αιτήσει εκθέσεις, άλλες εκθέσεις αυτών των ε, θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών κάναμε και μια σύντομη μελέτη. 12 θεσμικά όργανα, 41 υπηρεσίες και είχαμε 100% απαντήσεις. Ευτυχώς. Να προσθέσω επίσης ότι η έκθεση βιωσιμότητας δεν είναι μόνο έκθεση, αλλά και διαδικασία. Η έκθεση είναι το τελικό βήμα. Φυσικά Πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίζουν οι επιμέρους οργανισμοί και υπηρεσίε, τι είναι σημαντικό για εκείνους και μετά να χαράσουν μια στρατηγική. Επομένως, αναπόκειται ε, στον κάθε οργανισμό ε, να δει σε τι θα πρέπει να αναφέρει στην έκθεση και τι όχι. Λοιπόν, τα βασικά μηνύματα της επισκόπησης αυτής. Πρώτον, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη στρατηγική πέραν του 2020. Βέβαια, όταν αναφέρουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει, πρέπει να αναφέρουμε και τους στόχους. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι όλοι οι στόχοι και οι στρατηγικές έχουν να κάνουν μέχρι το 2020, ενώ το θεματολόγιο κινείται μέχρι το 2030. Πέρυσι, το Ελληνικό Συνέδριο είχε ήδη αναφέρει αυτό τον κίνδυνο ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αποφασίζεται χωρίς να υπάρχει ε, στρατηγική ευρύτερη τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση Κομισιών κατόπιν και συστηματικών εκκλήσεων ο πλευρά νομοθέτη. Τον Ιανουάριο υπήρξε λοιπόν ένα έγγραφο ανασκόπησης και αναστοχασμού ε, για με τίτλο «Προς ε, μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030». Όμως δεν είναι έκθεση βιωσιμότητας ούτε στρατηγική και δεν βρήκαμε κάποια ανάλυση για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση μα παρέπεψαν στην έκθεση τη Eurostat που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ε, περιγράφει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη βάσει στατιστικών δεδομένων από τα κρατη στην ουσία. Όμως και πάλι δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο συμβολής ε, του ενωσιακού προπολογισμού στην επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Είναι απλώ μια γενική περιγραφή. Τρίτον, σε ό,τι φορά την έκθεση επιδόσεων, θα περίμενε κανείς η Επιτροπή επίσης να υποβάλει έκθεση ως προς αυτό. Υπάρχει γενικά, υπάρχουν πολλές εκθέσεις επιδόσεων και δείκτες και το καθεξής, αλλά όλα αυτά δεν έχουν ε, ε, ενοποιηθεί υπό το πρίσμα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και ούτε υπάρχει εδώ η συμβολή του ενωσιακού προπολογισμού και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια. Προς ενημέρωσή σας μπορώ να πω ότι αυτό αντανακλά και το γεγονός ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μια στρεβλωμένη ε, αντίληψη ότι αυτοί οι στόχοι δεν αφορούν την Ευρώπη, αλλά τις μακρινές χώρες. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, μιλήσαμε και είχαμε επαφή με 12 θεσμικά όργανα και 41 υπηρεσίες. Ε, δύο ευρωπαϊκοί φορείς ε, δημοσιοποιούν έκθεση βιωσιμότητας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Συλλέξαμε και πληροφορίες, μάλλον και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες και κάποια να τα δημοσιοποιούν, στοιχεία, αλλά δεν είναι πλήρη αυτά τα στοιχεία, είναι αρκετά αποσπασματικά και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση των εργασιών και όχι στη στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην καλύπτονται σημαντικοί κίνδυνοι. Κλείνοντα λοιπόν, δεν υπάρχει υποβολή έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από, από του 43 φορεί που προανέφερα, μόλι δύο έχουν εκθέσει βιωσιμότητα. Και όπως προηγουμένως, η έκθεση είναι το τελικό βήμα μιας διαδικασίας και πολλές από τις προϋποθέσεις υποβολής τη έκθεσης δεν υπάρχουν. Πρέπει να έχει κάνει κάποιος να έχει χαράξει μια στρατηγική, να έχει κάνει την ανάλυση και βέβαια οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στον προπολογισμό και σε άλλες ουσιώδεις διαδικασίες για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε μια τέτοια έκθεση. Για το μέλλον λοιπόν έχουμε τέσσερις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή στρατηγική μετά το 2020 που θα καλύπτει τους, ε, τη βιωσιμότητα και τους σχετικούς στόχους. Δεύτερον, να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα στον ενωσιακό προπολογισμό και στο πλαίσιο επίδοσης. Τρίτον, να αναπτύξουμε τις εκθέσεις βιωσιμότητας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πέραν της Επιτροπής. Και τέταρτον, να αυξήσουμε την αξιοπιστία ε, των εκθέσεων μέσω των ελέγχων. Είναι σημαντικό αυτά τα φυλάδια να είναι μεν ευανάγνωστα, αλλά να έχουν και αξιόπιστα στοιχεία. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως δεν ήταν ε, ε, ε, πρόκειται για μια ε, σύντομη γενική έκθεση για την οποία είναι υπεύθυνη η συγκήτρια η συνάδελφος Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και ζητώ συγγνώμη που σας έχω γυρισμένη την πλάτη εδώ που κάθομαι. Βέβαια, διαβάζοντας ε, την ε, έκθεση αυτή, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει να θέσουμε ε, σε πράξη αυτά τα οποία διακηρύσσομαι και θα πρέπει να δούμε ακριβώς αυτά που εφαρμόζουμε και τις πράξεις μας ως υπηρεσίες, ως οργανισμοί, ως ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε πώς πρέπει να λειτουργούν οι όμιλοι, οι επιχειρήσεις όσον αφορά την βιωσιμότητα, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν ε, παίζουμε ρόλο. Ε, ορισμένες ε, υπηρεσίες ε, κάνουν αυτό το reporting, αλλά υπάρχουν δύο που αναφέρονται σε πιο υλικά ζητήματα και πώς μπορούν μέσω της χρηματοδότησης των προγραμμάτων να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όσον αφορά τη χρήση του ε, νερού, την χρήση του χαρτιού κλπ. Ε, οδηγούμε λοιπόν σιγά σιγά σε κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι η πιο σημαντική ε, πρέπει να αποτανθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι εδώ ακόμα η εκπρόσωπη της Κομισιόν, αυτό είναι καλό. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι θα πρέπει να ηγηθούμε δια του παραδείγματος. Φαντάζομαι ότι η απάντηση θα είναι ε, καταφατική, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα υλοποιήσουμε δηλαδή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, και πώς η Κομισιόν μπορεί να έχει μία πιο γενική στρατηγική επί αυτών των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε ε, αυτά που κηρύττουμε. Δεύτερον, πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, πρέπει να εισαχθεί νέα νομοθεσία. Μήπως θα πρέπει να διευρύνουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό. Και άλλη μία ερώτηση προς το ελεγκτικό συνέδριο η ερώτησή μου είναι, φαντάζομαι ότι περιμένετε λίγο ακόμα για να έχετε περισσότερα στοιχεία. Ωστόσο, ε, πιστεύετε ότι οι διαδικασίες απαλλαγής ε, του ε, Κοινοβουλίου είναι σωστές σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Λάρα. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Η Κομισιόν έχει δεσπίσει μεθοδολογία Είναι μία από τις ε, λίγες, από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς, ε, ε, τα λίγα θεσμικά όργανα που έχει πιστοτική γραμμή για, για το κλίμα. Βεβαίως αυτή η μεθοδολογία τελεί υπό αναθεώρηση. Ε, και ε, όταν θα υπάρχει η τελική εκδοχή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, θα ευθυγραμμιστεί και η μεθοδολογία. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πού βρίσκεστε όσον αφορά αυτή την αναθεώρηση της μεθοδολογίας. Επίσης, έχετε επισημάνει κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, γιατί όντως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές που αφορούν τεχνολογίες του κλίματος που όμως δεν καλύπτονται από τη μεθοδολογία της Κομισιόν. Βλέπω όμως αντίθετα ότι στην μεθοδολογία της Κομισιόν ιδιαιτέρως αντιπροσωπευτικό είναι το πρασίνισμα. Όμως από αυτά που λέει και το ελεγκτικό συνέδριο το πρασίνισμα έχει περιορισμένη, ε, περιορισμένο αντίκτυπο, περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Πού βρίσκεστε λοιπόν όσον αφορά αυτήν την αναθεώρηση της μεθοδολογίας έτσι ώστε να αξιολογήσετε κατά κάποιο τρόπο σωστά το τελικό προϊόν, να το ονομάσουμε έτσι. Ακόμα μια ερώτηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ε, χωρίς ε, να ε, προκύψει ε, πληθώρα διοικητικών ε, ρυθμίσεων ή διαδικασιών. Πρέπει με τον απλούστερο τρόπο να καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και μάλιστα τα αποτελέσματα να είναι αναλογικά προς το διοικητικό βάρος. Ολιβιέ Σαστέλ, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σημερίζομαι ε, ιδιαιτέρως ε, την ε, διαπίστωση της εισηγητρίας. Βλέπουμε μάλιστα και την ε, πολύ προχωρημένη εργασία του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την βιωσιμότητα και διαπιστώνουμε ότι η βιωσιμότητα δεν λαμβάνεται υπόψη στην, ανάλογη, στην, στον ελεγχοεπιδόσεων της Κομισιόν και μάλιστα δημοσιεύονται ε, διάφορες εκθέσεις ε, για την βιωσιμότητα. Είναι πολύ σημαντική η πρόκληση, κεφαλαιόδου σημασίας μάλιστα, που πρέπει χωρίς ε, ε, καθυστέρηση να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί βλέπουμε ότι με ορίζοντα το 2030 έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά ε, την βιωσιμότητα. Πότε θα έχει, μπορεί να μας πει η Κομισιόν, σταφή στρατηγική και όσον αφορά την περίοδο 2020-2030, πώς θα επιτύχει την βιωσιμότητα, πώς θα ελέγξει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Νομίζω ότι αυτά είναι ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα από την ανάγνωση αυτής της ε, έκθεσης. Ε, θα πρέπει να επαγρυπνούμε έτσι ώστε σε όλα τα θεσμικά μας όργανα, σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις υπηρεσίες ε, να ζητούμε να εντάσσεται αυτή η συλλογική, συνολική στρατηγική για την βιωσιμότητα σε όλα τα project και σε όλες τις πολιτικές. Και όχι να περιοριστούμε μονάχα στην μειωμένη χρήση ας πούμε χαρτιού ή νερού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε συγκεκριμένους στόχους ε, για το θέμα αυτό και να αναπτύξουμε καλύτερες πρακτικές, να ε, ε, οδηγήσουμε δια του παραδείγματος και οπωσδήποτε θα πρέπει να προσανατολίσουμε διαφορετικά κάποιους πόρους εκεί όπου η ευρωπαϊκή υπεραξία είναι απαραίτητη και εκεί που η βελτίωση είναι απαραίτητη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ η Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο ε, και την κυρία που μας έκανε την παρουσίαση καθώς επίσης και ε, τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κατέδειξε τις μη συμμορφώσεις που ε, προκύπτουν εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν προετοιμάζει ε, προϋπολογισμό και πι δελτα πι χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική για αυτά τα θέματα. Πώς είναι δυνατόν. Αυτό θα ήταν αδύνατον ε, σε μια επιχείρηση, δηλαδή αν δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Σας ευχαριστούμε που τα παρουσιάσατε όλα αυτά. Μία ερώτηση το ελεγκτικό συνέδριο έχει στοιχεία, εργαλεία, μηχανισμούς ε, πίεσης ε, ε, όσον αφορά το μέλλον. Έχει λοιπόν τα, τους μηχανισμούς, τα εργαλεία ε, αυτά που θα τις επιτρέψουν να πιέσουν την Κομισιόν, να την σπρώξουν κατά κάποιο τρόπο την Κομισιόν έτσι ώστε να προετοιμάζει ε, τα έγγραφα με, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχετε τέτοιους μηχανισμούς και εργαλεία στη διάθεσή σας. Όταν παρουσιάστηκε το πι και επιμείνατε ε, σε κάποια σημεία. Επί Πού βασιστήκατε μάλλον έτσι ώστε να κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις. Έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις ε, για την Κομισιόν όσον αφορά την 1η Νοεμβρίου ας πούμε. Θα τα καταφέρετε να καθορίσετε στρατηγική για τον προϋπολογισμό γιατί διαφορετικά δεν θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί τη κυρία Γκραπίνη ε, τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. Εναπόκειται σε εσά ε, πώς μπορεί κανείς ε, τους αριθμούς να τους εξηγήσει και ίσως μπορείτε και να μας δώσετε και μια καλύτερη γενική εικόνα. Μια εικόνα που να μην είναι γραφειοκρατική και να είναι προσαρμοσμένη σε όλες τις απαιτήσει. Αυτό είναι το καθήκον σας. Δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί κανείς να τα πει σε μία ξένη γλώσσα. Ε, θέλω μόνο να πω ότι όλα αυτά τα οποία έχετε να μας παρουσιάσετε είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Thank you, Ευχαριστώ ε, πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είναι δύσκολη ε, η θέση μου εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνετε στην Κομισιόν τη δυνατότητα να εξηγήσει την ε, θέση της. Φαντάζομαι ότι έχετε δει ότι σε αυτή την ε, περίπτωση του report δεν περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση της του συνεδρίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Λίνστρομ για αυτήν την έκθεση, γιατί η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκο. Η κυρία Λίνστρομ τα κατάφερε να ε, ε, συγκεράσει παλαιές πληροφορίες και στοιχεία με νέα στοιχεία. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά για την Κομισιόν στην προετοιμασία ε, της ε, επόμενης έκθεσης για την βιωσιμότητα. Φαντάζομαι όμως ότι μπορείτε να συμφωνήσετε. Το θέμα της βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ίσως είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς τα πράγματα, αλλά δύσκολο να τα υλοποιήσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, όταν επικοινωνούμε τα αποτελέσματα, να είμαστε σαφείς γιατί και τι ε, ε, επικοινωνούμε και επί ποιου ε, αναφερόμαστε. Ε, παρότι παρουσιάζεται η Κομισιόν ως, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, υπάρχουν μεμονωμένοι οργανισμοί, υπηρεσίες και η Κομισιόν είναι ένα από τα όργανα. Το reporting μπορεί να γίνει και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η κυρία Λίστρομα εξήγησε την ε, θέση της ε, ε, δημοσίου έναντι ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολύ περίεργες και περίπλοκες δομές. Για να εξηγήσουμε αυτά που κάνει η Κομισιόν, να πω ότι θα ήθελα να παραθέσω αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις ε, ε, που οδήγησαν στην ε, έγκριση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό που καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως δεσμευμένη όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, και βεβαίως θέλουμε να καλύψουμε όλους τους στόχους ε, μέσω σημαντικής ε, συμβολής και στην εφαρμογή του υλοποίησή τους και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι το monitoring, είναι, η παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ισχυρές αξιολογήσεις όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των στόχων. Ε, έχουμε διάφορα, ε, ε, διάφορους πυλώνες. Πρώτος είναι αυτός που αναφέρθηκε ήδη από την εισηγήτρια και είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, το report, στο οποίο βλέπουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει όσον αφορά ε, τους στόχους αυτούς στο σύνολό της και όχι ως, μεμονωμένες, ε, ε, ως μεμονωμένοι οργανισμοί. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έκθεση μπορεί κανείς να δει στοιχεία όσον αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσον αφορά μεμονωμένες χώρες και όσον αφορά κάθε έναν από τους στόχους. Δεύτερον, είναι μια έκθεση η οποία εγκρίθηκε για πρώτη φορά φέτος που ονομάζεται ε, ε, Σύνθεση report όσον αφορά την ε, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Εγκρίθηκε, παρουσιάστηκε μάλλον τον προηγούμενο Μάιο και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες συμμετέχουν στην υλοποίηση του στόχου της, του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής, του, των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Ε, ε, τρίτον, ε, είναι οι ίδιοι οι στόχοι και πώς τους παρουσιάζει ένα φόρουμ στο οποίο η Κομισιόν παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικός, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι ένα από τα στοιχεία επί των οποίων επέμεινε η κυρία Λίνστρομ. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε πληροφορίες για τα θέματα αυτά, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συμβάλλει ο προϋπολογισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στην απόκτηση επιπλέον επιπτώσεων. Αν δει κανεί τα παραρτήματα του προϋπολογισμού, θα ε, δει τις πραγματικές δηλώσεις όπου εξηγούνται ε, το πώς συμβάλλουν τα διάφορα προγράμματα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Προς ώρας ε, έχουμε ποιοτικές ε, πληροφορίες και θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμα, να δώσουμε ε, πληροφορίες σχετικά με όλες τις γραμμές του, προϋπο... του προϋπολογισμού έτσι ώστε να δώσουμε και στην Επιτροπή σας όσο γίνεται πιο σωστές πληροφορίες. Βεβαίως η Κομισιόν προσπαθεί να δει ε, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να βελτιωθεί για το μέλλον. Η Πρόεδρος Ούρσουλα Φοντερ θεωρεί ότι αυτά τα θέματα είναι από τις προτεραιότητες Βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε και βιώσιμη ε, Ευρώπη. Η Κομισιόν έχει ταυτοποιήσει τρία βήματα ε, και ε, τρία στοιχεία. Τα δύο έχουν ξεκινήσει, το άλλο πρέπει να υλοποιηθεί. Πρώτον, ότι η βιωσιμότητα είναι mainstream σε όλες τις στρατηγικές μας, πολιτικές μας. Ε, ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι mainstream σε όλες τις ε, πολιτικές και σε όλα τα προγράμματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πρέπει ε, να επιτηρούμε, να, παρατηρούμε την ε, προόδο και να είμαστε βέβαιοι ότι η πρόοδος αυτή είναι, είναι σωστή. Η Κομισιόν προτίθεται να βελτιώσει την ορατότητα της ετήσιας έκθεσης κατά την έννοια αυτή το τρίτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει ε, να ε, υλοποιήσουμε ε, είναι το εξή. Ε, η νέα πρόεδρος αναφέρθηκε στην βελτίωση, στην αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το εξάμεινο είναι ένα από τα κύρια ε, εργαλεία που έχουμε για τον οικονομικό συντονισμό. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις πρωτοβουλίε της νέας Προέδρου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορείτε να κατανοήσετε ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια μεταβατική φάση. Έχουμε το ΠΔΠ το οποίο συζητιέται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το, η τελική έκβαση αυτής της συζήτησης ε, θα μας δώσει την δυνατότητα να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα, ε, ε, ο, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μεταβατική ε, φάση, ότι είμαστε δεσμευμένοι όσον αφορά την βιωσιμότητα, ότι λαμβάνουμε πολλές αποφάσεις, αλλά πρέπει να περιμένουμε να ε, ε, ξεκινήσει πραγματικά η νέα Επιτροπή, έτσι ώστε όλες αυτές οι διαφορετικές ψηφίδες να μπουν στη θέση τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, μήπως ε, θέλει η συνάδελφος ε, Βόλτες να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να... Όχι, όχι, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ ήθελα να σας ε, ρωτήσω μόνο στη συγγήτρια αν έχετε κάτι να ρωτήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόντστρομ και θέλω να ρωτήσω την κυρία Λόντστρομ ε, στην δική της ε, την περιπτωσιολογία δεν φαίνεται η, καθόλου η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το ερωτώ αυτό γιατί, ξέρετε, εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα θέματα του προϋπολογισμού. Σας ε, ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας ε, και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, ε, πρέπει να πούμε ότι η βιωσιμότητα είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τις απασχόλησε και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Πολλοί πολίτες ε, θέλουν να γνωρίζουν ε, πώς ακριβώς ε, συμβάλλει ο προϋπολογισμός, τα κονδύλια του προϋπολογισμού στην βιωσιμότητα γενικότερα, όχι μόνο στην βιωσιμότητα σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και στην οικονομική βιωσιμότητα. Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά κάποιες από τις ερωτήσεις κατά πόσον αυτό μπορεί να εντάσσεται και στην ε, δήλωση αξιοπιστίας. Νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι έχουμε εκθέσεις για τις οικονομικές επιδόσεις και ε, εκθέσεις ε, για τη βιωσιμότητα. Το δεύτερο πρέπει να έχει σχέση με το πρώτο να τίθενται οι στόχοι και νομίζω ότι οι στόχοι της χιλιετίας ε, δημιουργούν ένα πολύ ωραίο πλαίσιο. Αυτό το στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός από τους 17 στόχους υπάρχουν και άλλοι στόχοι οι οποίοι έχουν εγκριθεί. Ως εκ τούτου το θεματολόγιο του 2030 προσφέρει ένα πολύ καλό πλαίσιο για το πώς πρέπει να γίνονται οι αναφορές για τη συνεισφορά. Όχι μόνο για το πώς ε, τα διάφορα προγράμματα σχετίζονται με τους ε, στόχους της χιλιετίας, αλλά ε, και επίσης ε, το πώς ε, η συνεισφορά μπορεί να ικανοποιήσει αυτό το στόχο. Επίσης Πολλά άλλα θέματα έχουν σχέση με την μακροχρόνια στρατηγική. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής πρέπει κανείς να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια και για τους 17 στόχους. Όσον αφορά την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν κάνουμε μόνο την ετήσια έκθεση, ε, αλλά επίσης ε, γνωμοδοτούμε και καταθέτουμε και έγγραφα ενημέρωσης. Ε, εμείς καταθέσαμε ένα τέτοιο έγγραφο για τις προτάσεις μας σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και για τα έσοδα εγώ σχολίωσα τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο ασκούμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι και αυτό το έχουμε εντάξει στην ετήσια έκθεση και θα συνεχίσουμε και να το κάνουμε. Συμφωνώ απόλυτα με το ότι οι εκθέσεις για τους στόχους της χιλιετίας δεν πρέπει να δημιουργούν νέα γραφειοκρατία και πιστεύω ότι οι καλύτερες εκθέσεις, οι βελτιωμένες εκθέσεις ε, για τις οικονομικές επιδόσεις είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά είναι σημαντικό αν θέλουμε να γίνεται αναφορά για το πώς ακριβώς τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα από εκθέσεις για τις οικονομικές επιδόσεις και όχι σε ξεχωριστές εκθέσεις για τη βιωσιμότητα. Και όσον αφορά στη μεθοδολογία ε, και στις, ε, στις ε, γρήγορες μελέτες περιπτώσεων έχουμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σχέδιο της έκθεσης το καταθέτουμε στην Επιτροπή και ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά τα σχόλιά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ολοκληρώσει η συγγήτρια. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ικανοποιητικέ οι απαντήσεις και διευκρινήσεις που ακούσαμε. Και πολύ ενθαρρυντικά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τομείς εργασίας. Συστήνονται ή πρόκειται να συσταθούν. Βέβαια, ξεκολουθώ να πιστεύω ότι η συνολική σφαιρική στρατηγική είναι απαραίτητη. Χωρίς με τη στρατηγική υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Βέβαια, υπάρχει και πρόβλημα αν δημιουργηθεί στρατηγική να οδηγηθούμε τελικά σε αλληλεπικαλύψεις και σε περιττές προσπάθειες. Όμως νομίζω ότι χωρίς τη στρατηγική υπάρχει ο κίνδυνος η έκθεση αυτή να είναι μια απλή έκθεση παρακολούθησης. Ενώ για μένα η έκθεση είναι και ένα ε, εργαλείο διαχείρισης και διοίκησης. Λοιπόν, μόνο η στατικική με προβληματίζει προ το παρόν. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι σημαντικά και είναι σημαντικέ οι τρει πρωτοβουλίε που ανέφερε η Κομισιόν. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Λίνστρομ και ε, θα ήθελα να συνεχιστούν αυτέ οι προσπάθειε και αυτέ οι εκθέσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λίνστρομ, το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και την κυρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά που μας είπαν και θα ασχοληθούμε με όλα αυτά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 5 της ε, ημερήσιας διάταξης. Ε, ε, πρόκειται για μια ειδική έκθεση που αφορά την συμμετοχή των πελιτών. Είναι το σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Ανεμή Τούτλμπομ έχει συντάξει αυτή την έκθεση εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Uh, Αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε την ειδική μας έκθεση για την πρωτοβουλία Have Your Say, ε, δημόσιες διαβουλεύσεις ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με τους Ευρωπαίους πολίτες. Αρχικά θα ήθελα να σας εξηγήσουμε γιατί κάναμε αυτή τον έλεγχο και να σας παρουσιάσουμε και το πεδίο εφαρμογή, την προσέγγιση και μετά τα ευρήματα και τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί κάναμε αυτή τον έλεγχο. Στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να διαβουλεύεται με τους ε, πολίτες ε, σε όλους τους ευρωπαϊκούς τομείς. Με ευρείε διαβουλεύσεις λοιπόν, δίνοντας ε, στους πολίτες και άλλα διαφορετικά μέλη να συμβάλλουν. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης του 2001, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δηλώνει την προσήλωσή της ε, να έρχεται σε επαφή με του Ευρωπαίου πολίτε σε όλο το δημοκρατικό κύκλο για να αυξήσει την ε, νομιμοποίηση και λογοδοσία στη νομοθετική διαδικασία. Παραπέμπουμε και στην στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2018-2020, όπου εντοπίζουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και θεσμικών οργάνων ως απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είμαστε μόνο θεματοφύλακε ε, των ε, οικονομικών συμφερόντων του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και συνήγοροι ε, του πολίτη. Και κλείνοντας υπάρχει και το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο του 2018. Το Κοινοβούλιο μας ζήτησε λοιπόν να αξιολογήσουμε πώς οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και κατά πόσο υπάρχουν ε, κατάλληλα και επαρκή εργαλεία διαφάνειας ε, και εξωστρέφειας. Τι ακριβώ εξετάσαμε. Θέλαμε να δούμε λοιπόν κατά πόσο είναι αποτελεσματικέ οι δημόσιε διαβουλεύσει ε, ό,τι αφορά την επαφή με του πολίτε και κατά πόσο αξιοποιούνται οι ε, συνεισφορέ του. Εξετάσαμε λοιπόν το σχεδιασμό του πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσο ανακλά βέλτιστε πρακτικέ, κατά πόσο η Κομισιόν διενήργησε τι ε, δημόσιε διαβουλεύσει με έναν τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά οι πολίτε να συμμετέχουν και κατά πόσο η Κομισιόν ανέλησε τα δεδομένα ε, και τι πληροφορίε που έλαβε με έναν ε, δημόσιο και διαφανή τρόπο. Κατά μέσο όρο, πάνω από 100 τέτοιε δημόσιε διαβουλεύσει γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί αναλύσαμε 26 που έλαβαν χώρα μεταξύ του 2006 και 2018 με πέντε γενικέ διευθύνσεις συνομιλήσαμε ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής, τη συνάφεια για τους πολιτες πολίτες συγγνώμη. Επισκεφθήκαμε δύο κράτη-μέλη και τον ΟΣΑ. Αναλύσαμε βασικά έγγραφα για τα ενδιαφέρουνα μέρη, τη συμμετοχή τους ε, και μιλήσαμε και με εμπειρογνώμονες για να βελτιώσουμε την ανάλυση μας. Έγινε και μια μελέτη αντίληψης με χιλιάδες ε, πολίτες που συμμετείχαν στα δείγματα ε, για τις δημόσιες για να συμπληρώσουμε τα ευρήματά μας και λάβαμε πάνω από 2.000 ε, απαντήσεις. Τι βρήκαμε λοιπόν. Και οι επιδόσεις του δείγματος και η αντίληψη ε, των πολιτών ήταν ε, αρκετά ικανοποιητική. 65% ήταν, δήλωσαν την ικανοποίηση ή μερική ικανοποίησή τους. Δεύτερον, εντοπίσαμε και τομεί ε, όπου μπορεί να υπάρξει βελτίωση στην διαδικασία δημόσιων διαβουλεύσεων. Αρχικά έχουμε χαμηλή συμμετοχή που εντοπίσαμε σε 26 δημόσιες διαβουλεύσεις στο, στο δείγμα μας. Το 1 τρίτο έλαβε κάτω των 75 απαντήσεων και μόλις ένα τρίτο έβαλε πάνω από χίλιες απαντήσεις. Και λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της Ευρώπης, είναι πολύ χαμηλός ε, ο αριθμός. Δεύτερον, ε, προβολή των δημοσίων διαβουλεύσεων. Είναι αρκετά περιορισμένη, βρήκαμε. Μόνο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ε, τα γνωρίζουν και πέραν της δημόσιας διαβούλευσης για ε, την θερινή και χειμερινή ώρα ε, που έτυχε δημόσιας προβολής, τα υπόλοιπα δεν ε, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω και άλλα τέτοια ζητήματα στις συστάσεις μας. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει μάλλον η εξαίρεση της ε, δημόσιας διαβούλευσης για την θερινή ώρα. Πέραν του, της, μάλλον παρά την υψηλή συμμετοχή, υπήρχε σημαντική γεωγραφική ανισορροπία. Οι περισσότερες απαντήσεις προήλθαν από τη Γερμανία, 3 εκατομμύρια περίπου, και την Αυστρία. Σε άλλα κράτη-μέλη, κυρίως στην Νότια και την Ανατολική Ευρώπη, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή σχεδόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντανακλάται στο σύνολο του δείγματό μα. Το 40% των απαντήσεων υπευλήθησαν την τελευταία ημέρα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Ήταν λοιπόν την τελευταία στιγμή όλα. Βελτίωση μπορεί να υπάρξει και στι διαδικασίε σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων, για την ασφάλεια δεδομένων και το feedback ε, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και τους ε, ε, κινδύνους. Δεν υπήρξαν συστηματικοί έλεγχοι κατά πόσο είναι αυθεντικές ε, οι απαντήσεις και ότι δεν ε, προκύπτουν από ρομπότ. Δεν ελέγχονται οι IP διευθύνσεις. Και απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι και συστήματα ασφαλείας για να μην υπάρχει χειραγώγηση των αποτελεσμάτων συστάσεις. Έχουμε έξι συστάσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει καλύτερα να παρακολουθεί τις δημόσιες διαβουλεύσεις, να βελτιώσει τις κατητήρες γραμμές του ευνομοθετήν με ειδικού δείκτες που θα πρέπει να παρακολουθούνται και να συμπεριλαμβάνονται σε εκθέσεις για όλες τις διαβουλεύσεις και συστηματικά να εξολογεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι των διαβουλεύσεων. Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσει η Κομισιόν τη στρατηγική της για τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Να εξηγήσει δηλαδή ποιες δραστηριότητες διαβουλεύσεων θα αξιοποιηθούν και πώς θα λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη, Ποιο είναι δηλαδή, ο σκοπός της δημόσιας διαβούλευση, διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρου, ε, λομπίστε, εταίρου άλλου, και να εξηγεί τον σκοπό και την ε, χρήση Καθώ και τη μετάφραση του περιεχομένου και των εγγράφων σε όλες τις γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, επιταχύνω λίγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει την εξωστρέφειά της, να προσαρμόσει τα μέτρα επικοινωνία και να έρχεται περισσότερη σε επαφή με τι ε, αντιπροσωπείε ε, στα κράτη-μέλη. Τέταρτον, το γλωσσικό ζήτημα και τα ερωτηματολόγια για να βοηθήσουμε τους πολίτες, όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν εύκολα και αποτελεσματικά, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τα κριτήρια για τις πρωτοβουλίες Εβραίου δημοσίου συμφέροντος, να μεταφράζει τα βασικά έγγραφα για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες ή τι πρωτοβουλίε Εβραίου δημοσίου συμφέροντο σε όλε τι επίσημε γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει ότι οι διαβουλεύσει γίνονται βάσει γενική μελέτη και δημοσκόπηση για το ευρύ κοινό. Μετά, επεξεργασία και ασφάλεια δεδομένων. Θα πρέπει να προστατεύονται οι δημοσιοβουλεύσεις κατά χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Αυτό θα γίνει με τον έλεγχο των ε, προτύπων που ακολουθούνται για την επεξεργασία δεδομένων και ε, να διασφαλίζει ότι οι απαντήσεις ε, την χάνουν σωστής σωστή Τέλος, αναδιάδραση, feedback προς τους, ε, τους πολίτες που έχουν δώσει απαντήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δίνετε τέτοιο feedback με διαφάνεια και εγκαίρος. Γιατί πολλές φορές είδαμε ότι απάντησαν πολίτες ε, στη δημοσιοδεβουλεύση, αλλά μετά τελικά δεν έμαθαν τι απέγιναν ε, οι παρατηρήσεις τους ε, ή τι έγινε τελικά με τη δημοσιοδιαβούλευση και να εξηγεί η Κομισιόν σε όσους απαντούν πώς έχουν ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις τους ή αν όχι γιατί δεν ελήφθησαν. Και με αυτές τις έξι συστάσεις καθίσταται σαφές ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των δημοσίων διαβουλεύσεων για να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή αυτή η γενική επισκόπηση. Ο συνάδελφο κύριο Πέξα είναι ο εισηγητή. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ελεγκτικό συνέδριο για αυτήν την ε, παρουσίαση. Ε, ε, όλα τα στοιχεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη με την πρόφαση ότι ε, υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ε, μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό στο μέλλον. Δεύτερον, είμαι περίεργος. Έχουμε όλα τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των χειρισμών Έχουμε κάνει αναλύσεις έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι ε, απαντήσεις οι οποίες ε, έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο αλλοιωθεί. Επίσης, έχουμε γενικούς αριθμούς σχετικά με το ποιο είναι το ποσοστό του Εβραίου κοινού που συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σε σύγκριση σχετικά με τους εκπροσώπους ας πούμε κλάδων, ε, οργανώσεων, οργανωμένων ε, ε, αντιπροσώπων κλπ. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω πώς είναι οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι απαντούν και μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται εδώ στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Τσίπολόνε από την Κομισιόν. Μάλλον είναι η κυρία Τσιπολώνε. Συγγνώμη που σας έκανα κύριο, κυρία, αγαπητή κυρία, αλλά θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ε, δυνατότητα να σχολιάσουμε την έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη μια τέτοια έκθεση και συμβάλλει στην βελτίωση της, ε, των διαδικασιών δημοσίας διαμούλευσης. Ε, θέλουμε να έχουμε ένα ρωμαλαίο σύστημα ε, διαβουλεύσεων και αυτό το αναγνωρίζει και το ε, κοινό και επομένως αυτό μας ε, εξασφαλίζει το γεγονός ότι έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης. Ε, βεβαίως το σύστημα διαβουλεύσεων λαμβάνεται υπόψη εις τις γενικότερες προετοιμασίες μας και συζητήσεις μας. Βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις ε, που, και στοιχεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Κυρίως ε, η σημασία του outreach, ε, δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να φτάσουμε σε όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα δουλεύουμε και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης το feedback, η ανάδραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, αλλά πάντα σε σεβασμό των ε, αρχών προστασίας δεδομένων στη διάρκεια της συλλογή των προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο εισηγητή, κυρίω όσον αφορά δε το θέμα της προστασίας των δεδομένων, έχω να πω το εξής. Η... Ε, συνήθως οι πολίτες απαντούν ε, κατανοώντας ότι τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν εντός ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και δίνουμε πάντα τον σύνδεσμο και υπάρχει η δυνατότητα για το ελεγκτικό συνέδριο να φτάσει στις 16.000 αυτές απαντήσεων. Επίσης, ε, ε, πρέπει στο μέλλον να ε, καταγράφεται σαφώς ότι μπορούν τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν και για έλεγχο που ενδεχομένως θα κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Στο μέλλον λοιπόν δεν θα υπάρξει το πρόβλημα αυτό. Επίσης υπάρχει μηχανισμός ταυτοποίησης. Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την διαβούλευση ε, να σας πω πάντως ότι ε, υπάρχει ε, αποκλισμός οποιος, οποιονδήποτε εξωγενών παραγόντων θα προσπαθήσουν να παρεμβληθούν έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Άρα, από τη μία μεριά θέλουμε περισσότερο outreach και από την άλλη πλευρά θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. αλλά ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένως θα είναι υπερβολικά ασφαλές ίσως δεν θα μπορεί να ε, ε, φτάσει στους πολίτες και να χρησιμοποιηθεί από αυτούς. Θέλουμε ε, γι' αυτό λοιπόν να μελετήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες χειρισμού ενδεχομένως και αλλίωσης των αποτελεσμάτων. Είμαστε όλες οι υπηρεσίες πολύ προσεκτικές όσον αφορά το θέμα αυτό. Όσον αφορά να σας πω ότι 80% των ε, απαντώντων είναι, και των συμμετεχόντων είναι απλοί πολίτες ε, το ευρύ κοινό είναι αυτό το οποίο στη μεγάλη πλειοψηφία συμμετέχει σε τέτοιες ε, διαδικασίες ε, διαβούλευσης. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι ιδιαίτερα προσφυλής η δυνατότητα στους πολίτες, η δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Να σας πω ότι στα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει τέτραπλασιαστεί η συμμετοχή των πολιτών και οι απαντήσεις. Βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί ε, το, η κατάσταση, να βελτιωθούν οι αριθμοί. Πάντως ήδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια ακολουθήσαμε αυξητική πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η συγκήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση σχετικά με την προστασία ε, δεδομένων. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει το privacy statement, άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον, ε, έτσι ώστε, γιατί για μας η πρόσβαση στα δεδομένα, στα στοιχεία είναι θεμελιώδους σημασίας. Καμιά φορά υπάρχει μια ένταση με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά νομίζω ότι τώρα πια ε, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Χάσαμε λίγο χρόνο βέβαια στη διάρκεια της έκθεσης αυτής. Ε, και ε, από τη δική μας, να σας πω ότι από τη δική μας πλευρά εμείς έχουμε ε, βεβαίως ε, περιφρουρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία, αλλά η Κομισιόν είναι η κύρια υπεύθυνη και κατά τη δική μας άποψη η κατάσταση δεν ήταν ιδεώδης. Ε, η Κομισιόν έχει στείλει την ε, έρευνα και θα πρέπει να δούμε η, η, αίσθηση είναι διαφορετική όταν ένα email φτάνει από την Κομισιόν ή αν το email φτάνει από δική μας διεύθυνση του ελεκτικού συνεδρίου. Ε, δεύτερον, όσον αφορά το θέμα της αλλίωσης, εμείς δεν βρήκαμε ε, τεκμήρια τέτοιου είδους αλλίωσης. Ε, απλώς ε, είδαμε ότι οι διευθύνσεις IP ε, εντός και εκτός της Ευρώπης δεν ελέγχονται ή τουλάχιστον εμείς δεν λάβαμε τέτοια πληροφορία. Στην παράγραφο 84 βλέπετε ότι η Γενική Διεύθυνση Digit ε, έκανα κάποιους ελέγχους ε, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και μάλιστα αναφέρεται ότι είτε η Γενική Διευθυντή είτε άλλες διευθύνσεις από ό,τι φαίνεται δεν ε, έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους ε, έρευνες ούτε για το γεωεντοπισμό ας πούμε διευθύνσεων IP. Ε, επομένως, ακόμα πολλά μπορεί να βελτιωθούν όσον αφορά αυτή την τεχνική πλευρά. Ε, και από την ε, στιγμή που ε, έχουμε διαβουλεύσεις που απαντούν ας πούμε 4 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 4,6 συγκεκριμένα και μετά αυτά, αυτές οι απαντήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για την διαμόρφωση πολιτικών θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλα γίνονται σωστά. Τέλος, όσον αφορά την απέτηση απάντησης, όπως είπα και προηγουμένως, Εάν ε, υπολογίσετε 500 εκατομμύρια πολίτες, ε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί είναι τέτοιοι έτσι ώστε να μας οδηγήσουν ε, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για σημαντικό εργαλείο. Πρέπει να αυξηθεί η ορατότητα της Κομισιόν. Όμως δεν συγκρίναμε αυτούς που απήντησαν εδώ με ε, τις απαντήσεις στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να φανταστώ όμως ότι σε ορισμένες ε, διαδικασίες διαβούλευσης και θα ξαναδείξω εδώ ένα slide, μια διαφάνεια που είδατε ότι σε έχουν in ...εξαιτίας 27, well, Uh, uh, Έχουμε διάφορες διαβουλεύσεις που σε μερικές είναι 6, άλλες 20, 27, 30, 34 συμμετέχοντες. Πάντως σε γενικές ε, γραμμές νομίζω ότι η ανάλυση μας μπορεί να είναι καλό εργαλείο, αλλά ε, οδηγούμε εδώ στη δεύτερη μας σύσταση, δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιο εργαλείο χρησιμοποιεί κανείς και για κάποιο στόχο. Δηλαδή ποιο είναι για τους ε, εμπορευόμενους, ποιο είναι για τους ε, ε, λομπίστες, ποιο για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, ποιο για το outreach των πολιτών κλπ. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάντως ε, τα θέματα και στους πολίτες. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για αυτό το σκοπό και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο φτάνει προς τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα διασφαλίσει και το δημοκρατικό χαρακτήρα αλλά και την ευκρίνεια ε, του νομοθετικού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Τουρλιμπλουμ. Ε, νομίζω ότι αυτά που είπατε πραγματικά θα διευκρινίσουν περαιτέρω την κατάσταση και θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή. Κοιτάξτε, ε, έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή ε, του κοινού. Αν κατάλαβα καλά, Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα η Επιτροπή να μετρήσει επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί και ε, ίσως θα μπορούσε να αλλάξει το IP του μέσα από ένα δίκτυο ε, προσώπων. Δεν ξέρω, ε, υπάρχει κάποια ανάλυση δεδομένων να μπορείτε να εντοπίσετε κάποια πλαστή δραστηριότητα, τέτοιου είδους δραστηριότητα. Και δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να ελέγξετε αν είναι αντιπροσωπευτική η δημογραφική εικόνα όσων απαντούν ή υπάρχει κάποια μετατόπιση. Γιατί μπορώ να φανταστώ ότι όταν απευθυνόμαστε στους ανθρώπους των κοινωνικών δικτύων, αυτοί είναι περισσότερο νέοι, οι οποίοι ε, είναι κατά κύριο λόγο οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Και ε, γι' αυτό ε, υπάρχουν άλλοι που δεν εκπροσωπούνται, υποεκπροσωπούνται. Μιλάω κυρίως ε, για το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι οι πιο ηλικιωμένοι έχουν διαφορετική άποψη για τις ε, συνέπειες ε, στην υγεία της αλλαγής της θερινής ώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρώτα απ' όλα ε, να πω, να είμαι σαφής όσον αφορά τις ερωτήσεις που κάνατε. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές ε, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συμμετέχει διπλά σε μία έρευνα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει. Ε, τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς στην έκθεσή μας είναι ο αριθμός των ανθρώπων ε, που συμμετείχαν σε διάφορες δημόσιες διαβουλεύσεις. Γιατί βλέπω ότι υπήρχε μία διαβούλευση με 12 μετέχοντες. Θα μπορούσε μπορούσε να είναι ο ένας άνθρωπος 12 φορές. Ε, δεν έχουμε κάτι που να το καταδεικνύει αυτό, αλλά μπορεί να γίνει. Όσον αφορά το δημογραφικό στοιχείο, στην παράγραφο υπαριθμών 12 αναφέρουμε ότι αυτή δεν είναι η αντιπροσωπευτική άποψη των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, είναι βεβαίως πολίτες που ενδιαφέρονται σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το 40% των πολιτών απάντησε στα αγγλικά παρότι κατ' ουσίαν μόνο το 5% των πολιτών χρησιμοποιεί τα αγγλικά στην καθημερινή του ζωή. Άρα δηλαδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το κοινωνικονομικό υπόβαθρο των πολιτών γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Αλλά μπορεί κανείς να υποθέσει ότι κατά κύριο λόγο πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφερόμενους πολίτες ε, κυρίως στις διαβουλεύσεις ε, ή στις έρευνες που έχουμε πολύ περισμένο αριθμό ανθρώπων που συμμετέχουν. Ε, ούτε και προβλέπετε ε, αυτό το εργαλείο να εκλαμβάνεται ως ε, αντιπροσωπευτικό. Αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι για την ανάδραση ένας από τους στόχους είναι να ε, βελτιωθεί η διαδικασία νομοθεσίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κάποιοι πολίτες είπαν χαιρόμαστε που μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά, αφού την πούμε. Ως εκ τούτου, αν δεν ξέρει κανείς σε ποιο εργαλείο χρησιμοποιεί για ποιο στόχο, είναι και πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα feedback. Γιατί ε, το να ε, διαβουλευτεί κανείς με 12 πολίτες. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία ή όχι και τι θα γίνει με τους 400 εκατομμύρια υπόλοιπους. Είναι καλό εργαλείο και θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι καλό το εργαλείο και είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει αυτή την απόφαση, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στις δικές μας συστάσεις, ε, παραδείγματος χάρη σε μία σύσταση λέμε η γλώσσα. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον θα γίνει μετάφραση ε, στα αγγλικά ή και στις 24 ε, ευρωπαϊκές γλώσσες. Όμως δεν είναι απόλυτα σαφές ποιες έρευνες θα μεταφραστούν και ποιες όχι. Και έτσι απαντάω στην ερώτησή σας ποιο είναι το δημογραφικό υπόβαθρο. Κοιτάξτε, αν δεν γίνει μετάφραση σε όλες και στις 24 γλώσσες, τότε ορισμού αποκλείει κανείς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ε, όχι μόνο δεν είναι αγγλόφωνοι, αλλά δεν μπορούν καν να συνοηθούν στα αγγλικά. Ως εκ τούτου, αν δει κανείς ε, τις ε, έρευνες που φτάνουν σε πολλούς ανθρώπους, εκεί βλέπει κανείς ότι υπάρχει γεωγραφική ανισορροπία και πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί η ε, Γερμανία και η Αυστρία συμμετέχουν κυρίω και όχι οι χώρες χώρε ούτε του Νότου είτε της Ανατολικής Ευρώπης. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί κανεί ε, να πει ότι ε, οι άνθρωποι το θέλουν, άρα το κάνουμε. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε. Γι' αυτό λοιπόν στην σύσταση παρελθόν 2 λέμε ότι ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πει ότι χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για αυτό το στόχο, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι, πολύ, ε, θα είναι σαφέστερα. Έχω την εντύπωση ότι και η Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο. Yes. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι για το θέμα της ασφάλειας. Πρόκειται για διαδικτυακές διαβουλεύσεις. Και εμείς λοιπόν έχουμε πολύ υψηλά πρότυπα ασφαλείας, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να μπει στους ιστοτόπους μας, όχι πάντα για τους σκοπούς διαβούλευσης. Γι' αυτό οποτεδήποτε υπάρχει μία ανομαλία σε ό,τι φορά την ε, ε, χρήση, ε, πάντα αυτό γίνεται αντιληπτό και πάντα προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο στις εκστρατείες έχουμε πραγματικούς χρήστες και όχι πλαστές ε, διευθύνσεις IP που προκύπτουν από bot. Για τα δημογραφικά στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε. Ξέρουμε δηλαδή ε, οι συμμετέχοντες στη ηλικία είχαν κατά μέσο όρο και το καθεξής. Για παράδειγμα, κάποιες διαβουλεύσει ε, για το πρόγραμμα έρασμο. εκεί προφανώς είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον στους νέους, όμως ε, βλέπουμε ότι ανάλογα ε, με τον τύπο διαβούλευση, αλλάζει και η μορφή δημοσιοποίηση και τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιούμε. Τέλος, αυτή η διαβούλευση είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως υπόθηκε σωστά λοιπόν, δεν είναι αντιπροσωπευτικό μέσο, δεν είναι ε, δημοψήφισμα. Είναι όμως ένα μέσο που χρησιμοποιούμε και θέλουμε να δίνουμε και feedback προς τους πολίτες για να γνωρίζουν πώς ακριβώς αναλύσαμε τις απαντήσεις τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι ο εισηγητής κλείνοντα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο από μένα. Πολύ ωραία. Ως εκ τούτου διευκρινίσαμε κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τούτσι για όλα αυτά που μας είπε. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Και τώρα ο εισηγητής μας ίσως ε, μπορεί να προσπαθήσει να καταρτήσει ένα έγγραφο εργασίας. Αυτά. Λοιπόν, διακόπτουμε τη συνεδρίαση και στις 3 ε, η ώρα θα ξεκινήσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γι' αυτό παρακαλώ τους ε, συναδέλφους ε, να είναι παρόντες. 3 με 3 και 4 και μετά θα περάσουμε στην έκθεση Όλαφ με τον εισηγητή Μαρινέσκου. Γεια σας.